Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, σα καλωσορίζω στη συνεδρία τη Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού για σήμερα και για αύριο. Έχετε την ημερήσια διάταξη, δεν έχει δει κανεί αλλαγέ εξ όσων γνωρίζω. Όσοι μιλούν τώρα στην αίθουσα παρακαλούνται να μην μιλούν δυνατότερα εμού. Ε, γνωρίζετε την ημερήσια διάταξη, λοιπόν δεν χρειάζονται αλλαγέ, επιθυμίες, εν δεν έχουμε για τροποποίηση. Στο σημείο 2 να σα πω τι γλώσσε έχουμε, όπως πάντα μεταδιδόμαστε στο διαδίκτυο. Και πάμε στο τρίτο σημείο ήδη, που είναι η μελέτη για τα ε, μεγάλης κλίμακας έργα υποδομής και ε, διαδικασίες συμβάσεων. Ε, εισηγητής είναι ο κύριος Βάλλη και θα μας παρουσιάσουν ο κύριος Κάμπη και ο κύριος Άκερμαν από την Pro Mayer Sons. Ποιος θα αρχίσει πρώτος. Παρακαλώ, καλωσορίσατε και ε, με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε να ακούσουμε τη μελέτη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που έχουμε να σας παρουσιάσουμε τη μελέτη ε, σήμερα. Κανονικά, εγώ δεν θέλω να αρχίσω με περιορισμούς, αλλά θα πρέπει να τονίσουμε ότι κατεβλήθη μια προσπάθεια να δώσουμε γενικές κατευθυντήριες γραμμές και κάποιες πολύ γενικές συστάσεις για τα όσα συμβαίνουν. Τούτο λοιπόν λεχθέντων θα σας παρουσιάσουμε κάποιες διαφάνειες που καλύπτουν και το πλαίσιο της ε, μελέτης, τα βασικά ευρήματα και κάποιες συστάσεις που θα θέλαμε να ε, σας απευθύνουμε σε ό,τι αφορά το πλαίσιο. Ποια ήταν η ιδέα της μελέτης να ε, κατανοήσουμε καλύτερα, έχοντας προετοιμαστεί, ε, την εμπειρία που συνδέεται ακριβώς με την προετοιμασία και την σύναψη συμβάσεων για έργα υποδομών μεγάλης κλίμακας που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το ΕΦΣΥ και την διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Αυτές είναι οι τέσσερις χρηματοδοτικές πηγές. Έχει σημασία να τονίσουμε ότι σήμερα Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση 14% του ΑΕΠ ε, κινείται μέσω δημοσίων συμβάσεων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και 50% των κονδυλίων ε, ΕΣΥΦ ε, διακινούνται μέσω δημοσίων συμβάσεων. Επίσης, άλλο σημαντικό που πρέπει να συγκρατήσουμε ότι 13 κράτη-μέλη, σύμφωνα ε, με το αντίστοιχο βαθμολόγιο της εσωτερικής αγοράς για τις ε, δημόσιες προμήθειες, χωλένουν 13 κράτη-μέλη. Είναι κάτω από τη βάση βαθμολογία τους, μάλλον αρνητική και όχι ικανοποιητική καλή. Αυτά θα τα δείτε στη σελίδα 25 της μελέτης ε, που θα λάβετε σε μια γραφική παράσταση. Το Ευρωπαϊκό Λεκτικό Συνέδριο το 2017 ετώνησε ε, τον τρόπο με τον οποίο ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός προστατεύεται στις διάφορες πρακτικές συμβάσεων ε, των ευρωπαϊκών κρατών μελών. Στην έκθεση του ΔΕΓΙΑ το 2016 ετώνησε ότι υπάρχουν κάποιοι τομείς όπου χωράει βελτίωση ε, και αυτά τα λέει η μελέτη ε, πολύ σύντομα όμως σας τα δείχνουμε στο, στην διαφάνεια και ε, στις οθόνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν χωράει πάντα βελτίωση και για την προετοιμασία και στην εκ των προτέρων αξιολόγηση. Υπάρχουν και κάποιες διοικητικές καθυστερήσεις που είναι κοινή πρακτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, επίσης κάποια προβλήματα και περιορισμοί στις ικανότητες και δυνατότητες που έχουν οι ομάδες που προετοιμάζουν τους φακέλους. Αυτά λέγει ε, η έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου το 2016 και θα ήθελα να τα υποβάλλω υπόψη σας. Στη σελίδα 25 της μελέτης βλέπετε αυτή τη γραφική παράσταση που εμφανίζεται και στις οθόνες και βλέπουμε ότι ε, υπάρχει σημαντικό μέρος ε, τμήμα των κρατών μελών 13, όχι η πλειονότητα, αλλά που υπολείπονται ενό ελάχιστου κατοφλίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό Λοιπόν, η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για μεγάλα έργα υποδομής στις σημερινές δημοσιονομικές προπτικές είναι 120 δισεκατομμύρια. Εδώ βλέπετε την κατανομή ανα, ε, μέσω χρηματοδοτικό από τα τέσσερα που σας είπα προηγουμένως. Και επίσης ε, θεωρήσαμε ενδιαφέρον να δούμε πώς επενδύουν τα κράτη-μέλη στις υποδομές ενέργειας και μεταφορών που είναι και αυτή πολύ ωραία γραφική παράσταση και βλέπετε τη σημασία που έχουν αυτές ε, οι επενδύσεις. Και αφορά και τα κράτη που μπήκαν το 2004, το 2007 και πιο πρόσφατα η Κρότια. The uh, Η μελέτη προφανώς καλύπτει τις πρακτικές όλων των κρατών μελών και καταλαβαίνετε ότι είναι 3.000 σελίδες. Ουσιαστικά 100 σελίδες θα χρειαζόμασταν ανά κράτος μέλος και μετά για να τονίσουμε τις βασικές τάσεις θα θέλαμε και άλλες τόσες σελίδες. Γι' αυτό είχαμε κάποιο περιορισμό. Παρ' όλα αυτά έχουμε κάνει λεπτομερή ανάλυση σε τέσσερις χώρες. Τσεχική Δημοκρατία, Ισπανία, Ελλάδα και Ρουμανία. Και θα βρείτε τα συμπεράσματα μας στη μελέτη σε μεγαλύτερες λεπτομέρειες και υπάρχουν και τέσσερις χώρες ε, όπου έχουμε μελετήσει τέσσερα συγκεκριμένα έργα. Το ένα είναι διασυνοριακό και ήταν ένα έργο πολύ ψηλά στην πολιτική, ε, στις πολιτικές προτεραιότητες. Ε, η συνδρομική σύνθεση Λιών Τωρίνου επίσης ε, αυτοκινητόδρομο στην Ολλανδία, στην Κύπρο και ε, ε, τα έργα για την ανακαίνιση της γραμμής 5 στο μετρό της Μαδρίτης. Αυτά είναι τα σημαντικότερα στοιχεία που διακυβεύονται. ποια ήταν τα ευρήματα. Το σημαντικό είναι να ε, γνωρίσουμε ποιος κάνει τι ε, σε αυτή την υπόθεση. Τα κράτη-μέλη καταρτίζουν τους φακέλους και εκτελούν το έργο. Ε, κάνουν την περισσότερη δουλειά, απλά λόγια. Και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί ε, καλούνται να ελέγχουν τη συμμόρφωση. Άρα οι περιορισμοί έχουν να κάνουν με τις περιορισμένες δυνατότητες και ικανότητες που έχουν τα κράτη-μέλη, γιατί είναι λίγοι υπάλληλοι που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, τα οποία είναι πάρα πολύ περίπλοκα και χρειάζονται πολύ ισχυρή κατάρτιση και γνώσει και προσόντα που αποκτά κανεί με το χρόνο. Και επίση, σε αυτή την περίπτωση ένα περιορισμό που έχουμε ε, ανακαλύψει και λάβει υπόψη μας καθ' όλη τη διάρκεια της μελέτης. Γενικώ λοιπόν ε, η ε, γνώμη των εμπειρογνωμόνων λέγει ότι όταν πρόκειται για αξιολογήσεις εκ των προτέρων, μελέτες αντικτύπου, αναλύσεις κοινωνικο-οικονομικές και κόστους ωφελίας, ε, είναι σωστή, καλή η πρακτική, ικανοποιητική. Μπορεί να είναι αυτό πολύ γενικό λόγο και αφηρημένο. Πάντα θα βρούμε ε, κάποιο αρνητικό ε, παράδειγμα ή αρνητική πρακτική, αλλά γενικά είναι ικανοποιητικά. Φυσικά πάντα χωράει βελτίωση και θα θέλαμε και εδώ να τονίσουμε κάποια στοιχεία. Πρώτον, τα περιβαλλοντικά θέματα. Δεύτερον, η σημασία που έχει κανείς να εξετάζει τις παρεμβάσεις ε, ως προς τις επιπτώσεις του. Δηλαδή όταν φτιάχνεις ένα κομμάτι αυτοκινητοδρόμου, τι θα σημαίνει αυτό για την ευρύτερη περιοχή ε, και τι τόπο θα πιάσουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια στην ευρύτερη περιφέρεια και χωράει η βελτίωση. Ε, η διαφάνεια στην κατάρτιση του φακέλου επίση θα μπορούσε να βελτιωθεί κατά τη γνώμη μας και επίσης βρήκαμε ότι δεν συμμετέχουν πάντα όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Γίνεται μια διαβούλευση, ας πούμε, αλλά με την κοινωνία των πολιτών και τους πολίτες δεν είναι πάντα η καλύτερη δυνατή επιθυμητή. Το ξέρω ότι είναι γενικά σχόλια αυτά, αλλά επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, είναι περιορισμένος ο χρόνος, θα ήθελα να επικεντρωθώ σε αυτά τα βασικά. Εδώ λοιπόν θα δείτε και άλλες ε, γραφικές παραστάσεις και σχεδιαγράμματα που δείχνουν ποια είναι η κλασική κατανομή των ρόλων ανάμεσα στα κράτη-μέλη και ε, τα χρηματοδοτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τους ενδιαφερομένους. Εδώ σας έχω ε, στην οθόνη την περίπτωση του ΕΦΣΙ, του τραμίου Στρατηγικών Επενδύσεων. Για άλλα ευρήματα τώρα στην επόμενη φάση της υπογραφής της σύμβασης, όχι στην κατάρτιση του φακέλου. Σήμερα τουλάχιστον δεν έχουμε ε, αρκετή γνώση για το τι συνέβη με τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα θέματα που σας παρουσιάζω σήμερα. Δηλαδή, ε, προαιρετική ε, αξιολόγηση εκ των προτέρων, ε, να γίνουν πιο επαγγελματικές οι δημόσιες συμβάσεις και να υπάρχει καθοδήγηση για τις δημόσιες συμβάσεις. Δεν ξέρουμε τι συνέχεια έχει δοθεί σε αυτό, γι' αυτό θα έχει σημασία να αναλύσουμε η σημερινή απήχηση αυτών των ανακοινώσεων των συντομότερο δυνατών. Όπως σας είπα και προηγουμένως, γενικώ πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθούν ε, με ικανοποιητικό ε, τρόπο ε, όλα αυτά, αλλά και πάλι χωράει βελτίωση. Δεν αξιοποιείται πλήρως η δυνατότητα που προσφέρουν τα ίδια τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Υπάρχει απορρόφηση οι βέλτιστες πρακτικές, οι εμπειρίε, οι γνώσει είναι στη διάθεση των κρατών μελών. Αλλά είναι πάρα πολύ λίγα τα κράτη-μέλη τα οποία αξιοποιούν και χρησιμοποιούν αυτό το υλικό που τους ε, διαθέτουν τα θεσμικά όργανα. Για τη συλλογή δεδομένων θα μπούμε σε λεπτομέρειες αργότερα και εκεί χωράει μεγάλη βελτίωση. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν, γιατί πιστεύουμε ότι είναι σημαντικά όλα αυτά, διότι αυτό θα επέτρεπε μια εκ των υστέρων εξακρίβωση ε, κατά πόσο συμμορφώνεται το έργο με τους αρχικούς στόχους ε, ε, που περιλαμβάνει η σύμβαση. Ο συνάδελφος τώρα. Τι άλλο κοιτάξαμε. Το θέμα της ανάθεσης συμβάσεων με μία προσφορά ήταν σοβαρό πρόβλημα. Συμβάσεις που ανατίθεται άμα την παραλαβή μίας προσφοράς. χρησιμοποίησαμε στοιχεία που κατεβάσαμε από την πύλη ανοιχτών δεδομένων, ηλεκτρονικά στοιχεία για τους διαγωνισμούς, περίοδος 2009-2017. Τα στοιχεία δεν είναι πολύ αξιόπιστα. Θα έρθω σε αυτό σε λίγο. Ξεκινήσαμε με 4,6 ανακοινώσεις για τις συμβάσεις και λείπανε κάποια στοιχεία. Και είχαμε πολύ ψηλά ποσά, ασυνήθιστα υψηλά ποσά. Και είχαμε ανακοινώσεις για ανάθεση 240.000 διαγωνισμού με ποσά από 1 εκατομμύριο μέχρι ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Και τι είδαμε. βλέποντας όλους τους διαγωνισμούς που είχαν δημοσιευθεί ημερήσια, δηλαδή προμήθειες με πώς Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή χωρίς, περίπου 12% χρηματοδοτήσεως, που ανετίθετο, ανετίθετο με μοναδικές προσφορές, με μια και μοναδική προσφορά. Για έργα με χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ενώσεως, οι αριθμοί ήταν χαμηλότεροι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου 9% των συμβάσεων ανατέθησαν με βάση ε, μίας και μοναδικής προσφοράς κάθε σύμβαση. Βλέπετε το διάγραμμα. Με πιο ανοιχτό χρώμα βλέπετε τη χρηματοδότηση συνολικά και με Ευρωπαϊκή Ένωση και χωρίς Ευρωπαϊκή Ένωση, χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοτεινή, το σκοτεινό διάγραμμα δείχνει τις, ε, τους διαγωνισμούς με αποκλειστική χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Βλέπετε ότι η ανάθεση με μοναδική προσφορά ποικίλει από την περίοδο 2009 μέχρι το 2017. Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο όπου έχουμε σχέση με πόρους Ευρωπαϊκής Ενώσεως, το ποσοστό χρηματοδοτήσεως που εμπλέκεται με αναθέσεις με μια προσφορά είναι χαμηλότερο όταν εμπλέκεται η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ό,τι στις άλλες περιπτώσεις που δεν έχουν τέτοια περίπτωση. Λοιπόν, βλέποντας συνολικά τι έγινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξετάσαμε και τρεις συγκεκριμένες χώρες, Πολωνία, Ουγγαρία και Δανία. Και τι βλέπουμε στον πίνακα. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως βλέπουμε και στην πρώτη διαφάνεια, 12% των συμβάσεων αφορούσαν μία προσφορά και 9% ε, αφορούσαν μοναδική προσφορά με εμπλοκή των πόρων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην Πολωνία και Ουγγαρία. Το συνολικό ποσό της χρηματοδοτήσεως που ενεπλέκεται σε μοναδική προσφορά συνολικά ήταν πιο ψηλό για όλες τις συμβάσεις αλλά αρκετά χαμηλό σε περίπτωση εμπλοκή χρηματοδοτή Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Τι δείχνει ο πίνακα, όπου υπάρχουν άλλα κράτη-μέλη όπου αναθέσει μέσω μια προσφορά με εμπλοκή χρηματοδοτή Ευρωπαϊκή Ενώσεω είναι πιο ψηλό από ποσοστό των αναθέσεων. Στην Πολωνία και στην Ουγγαρία, πίνα. Στη Δανία Όταν έχουμε χρηματοδότηση τη ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ελάχιστη ανάθεση ε, με ε, μία προσφορά. Τι ανέφερα. Ανέφερα κάποια προβλήματα όσον αφορά τα στοιχεία που κατεβάσαμε από την πύλη με τα ελεύθερα στοιχεία. Περίπου 42% των αρχείων, 4,6 εκατομμύρια αρχεία δεν είχαν κάποιες κρίσιμες αξίες, όπως το ποσό της συμβάσεως που ανετέθη, κατά πόσο είχαν εμπλακεί χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωση. Έπρεπε αυτά τα στοιχεία να τα βγάλουμε εκτός, να τα αφήσουμε εκτός. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάποια ανάλυση. Κάτω από χίλια, χίλιες τέτοιες περιπτώσεις είχαμε όπου τα ποσά ήταν πάνω από ένα δις. Ίσως Υπάρχουν κάποιες αναθέσεις πάνω από ένα δις, οι δύο κάτω σειρές, η κάτω σειρά δείχνει την υψηλότερη τιμή. Πώς να το πω τώρα αυτόν τον αριθμό. Για το Υπουργείο Μεταφορών της Βουλγαρίας. Λοιπόν, η χώρα που είχε ε, πει αυτή την ε, σειρά ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο. Τι έγινε κατά τη διάρκεια της εισόδου των στοιχείων ή ε, επεξεργασίας των στοιχείων έγινε το μπέρδεμα. Βλέπουμε το παράδειγμα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε αναλύοντας τα στοιχεία. έχοντας αφήσει εκτός πολλές πληροφορίες, όπου είδαμε ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν έχουμε εμπιστοσύνη ότι έχουμε πολύ ακριβή στοιχεία. Ακόμα και για τα διαγράμματα και τους πίνακες που σας παρουσιάζουμε. Ποιο είναι το θέμα. Όπου η ηλεκτρονική αυτή διαγωνισμοί σχεδιάστηκαν διαφορετικούς σκοπούς και τα στοιχεία δεν ταιριάζουν αυτή την ανάλυση. Για να μπορούμε να διαπιστώσουμε εκ των υστέρων πώς η χρηματοδότηση έχει ανατεθεί, τι ποσά έχουν ανατεθεί και να κάνουμε την ανάλυση. Υπάρχει κενό. Στα στοιχεία. Παρόλο που η κατάσταση βελτιώθηκε. Πριν από κάποια χρόνια κάναμε παρόμοια ανάλυση. Τα διαθέσιμα στοιχεία απεκτήθησαν από το Open TED. Μαζεύτηκαν κάποιοι hackers για κάνα διήμερο, πήραν στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προσπάθησαν να τα επεξεργαστούν και τα δημοσιεύσουν. Αυτό που έχουμε εδώ αποτελεί τεράστια βελτίωση σε σχέση με αυτό. Αλλά, αλλά δεν είναι αξιόπιστα τα στοιχεία για τους σκοπούς που θέλαμε. Άλλα ευρήματα από τη μελέτη όσον αφορά την εξέταση αναχώρα. Συχνές αλλαγές του ρυθμιστικού πλαισίου. Περιορισμένος συντονισμός μεταξύ των αρμοδίων αρχών. Περιορισμοί χωρητικότητας δυνατοτήτων, το προανέφερα δίνεται αποκλειστική προσοχή στην τιμή περισσότερες φορές παρά στην ποιότητα της προσφοράς, τεχνητός διαχωρισμός των κονδυλίων των έργων σε λιγότερο από 10% των περιπτώσεων, αλλά εξακολουθεί να ισχύει και κάποια διαφθορά, ατασταλίες, τα γραφήματα σελίδες 29 και 31, κοιτάξτε, της έκθεσης. Βλέπετε τις ατασταλίες που έχουν τοπιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πολιτικής Συνοχής, σελίδα 31, έκθεση Όλαφ για τα σταλίες που, που επηρέασαν το ε, ESF πέρσι, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Περιορισμένος έλεγχος μπορεί να γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτό σχετίζεται και με τους περιορισμένους πόρους και δυναμικό. Ενώ ο ρόλος που πρέπει να διαδραματιστεί απαιτεί περισσότερους πόρους και στελέχωση. Για να μην μακρηγορώ, θα συγκεντρωθούμε τώρα στις συστάσεις μας προς εσάς σαν Επιτροπή. Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης. Πιστεύουμε καταρχάς ότι χρειάζεται συλλογή στοιχείων και καλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων που έχουν τα κράτη-μέλη όσον αφορά τις κρατικές προμήθειες κυρίως για έργα μεγάλης κλίμακας. Πρώτο συμπέρασμα αυτό. Δεύτερο, πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη κατανόηση του αντιχτύπου των διαφόρων πρωτοβουλειών που δρομολογήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα. Δεν θα τις αναφέρω εκ νέου, τις βλέπετε στην οθόνη. Πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει μια ανάλυση των λόγων για τους οποίους οι διαθέσιμοι πόροι που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη-μέλη δεν χρησιμοποιούνται. Υπάρχει τεχνογνωσία. Πολύ σπάνια χρησιμοποιείται τα κράτη-μέλη όμως. Και βάσει των όσων είπε ο συνάδελφος, χρειάζεται να δούμε τα κενά και τις ασυνέπειες που υπάρχουν στα στοιχεία. Διότι είναι μόνη βάση δεδομένων που έχουμε για ανάλυση. Και τέλος, εξίσου σημαντικό. Πιστεύουμε ότι σε κάθε διαδικασία διαγωνισμών πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο οι ενδιαφερόμενοι, οι σχετικοί. Σας ευχαριστώ. βλέπετε κάπως μπερδεμένοι, όσο πολύ μπερδεμένοι, γιατί έχουν τεράστια σημασία αυτά τα στοιχεία που μας δίνεται και που έχουν πολύ μεγάλη διαφορά από αυτά που μας έχουν δώσει από την, ε, Επιτροπή των, από την ε, Υπηρεσία Μελετών και από αυτά που έχουν δηλώσει τα κράτη, όπως Πολωνία, Κροατία, 45% των ευρωπαϊκών κονδυλίων ε, με συμμετοχή μόνο μίας επιχείρησης. Φαντάζομαι ότι έχετε μεγαλύτερη βάση δεδομένων σε θέση σας αλλά δεν νομίζω ότι θα άλλαζαν τόσο ριζικά τα στοιχεία. Άρα έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα ως προς τα δεδομένα πάνω στο οποίο στηριζόμαστε. Και τη ρωτώ με ποιο είναι το πρόβλημα ακριβώς. Ο κύριος Βάλιος, γιατί έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το θέμα των ε, στοιχείων Είναι όντω δύσκολο να αναλυθούν τα στοιχεία, όπω είπε και η, Πρόεδρο, στο θέμα των ε, μεγάλων υποδομών, των ε, κρατικών προμηθειών κτλ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάντω του ε, υπεύθυνου τη μελέτη που έκαναν πολύ μεγάλη δουλειά, πολύ σοβαρή δουλειά. Προσπαθούν να παρουσιάσουν και μια ανεξάρτητη θεώρηση και έναντι των θεσμικών οργάνων σε σχέση με τη διεξαγωγή αυτών των μεγάλων έργων υποδομών. Υπάρχουν στοιχεία λοιπόν στη μελέτη όπου αναλύονται οι διαδικασίε προετοιμασίας και διεξαγωγής των δημοσίων ε, προμηθειών. Και εδώ έχουμε ένα 14% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ ε, μεταξύ 14 και 20, ε, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί κατά 120 δισεκατομμύρια ευρώ τα έργα αυτά. Είναι τεράστια τα ποσά λοιπόν, οπωσδήποτε πρέπει να μεριμνούμε ώστε να χρησιμοποιούνται σωστά το ελεγκτικό συνέδριο, όπως και η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, έχουν εντοπίσει αρκετές αδυναμίες στην εκτέλεση και απορρόφηση των κονδυλίων. Αυτό άλλωστε το καταγράφουν και τα στοιχεία. Το επισημαίνει και η πρόοδος ότι είναι δύσκολο κάπως να βρούμε τι, τα σωστά στοιχεία, ή μαρλού τις σωστές αντιστοιχίες στη μελέτη και ιδιαίτερα σε σχέση με τις εκ των προτέρων αξιολογήσεις της πραγματικής προστιθέμενης αξίας. Βλέπουμε ότι πολύ συχνά αυτές, οι εκ των προτέρων δηλαδή αξιολογήσεις, βρίσκονται σε μια δυσκολία γιατί υπάρχουν κάποιες, κάποιες ε, περιπτώσεις που χρειάζονται πολύ περισσότερη προσοχή ώστε να μην, τεθούν και, να μην τεθεί και η ανεξαρτησία αυτών των μελετών. Οι εξάντε λοιπόν αξιολογήσεις ε, δεν πρέπει να υποτάσσονται σε πολιτική βούληση ή προτίμηση. Η αξιολόγηση λοιπόν και κυρίως περιβολητικού χαρακτήρα έχει γίνει κατά τρόπο ανεπαρκή, αδύναμο ή ε, κακό χρειάζονται βελτιώσεις ώστε να εξασφαλιστεί πως όλες οι πτυχές της αξιολόγησης ε, αναπτύσσονται πλήρως για να αποφευθούν και τα σφάλματα του παρελθόντος, αυτά που έχουμε εντοπίσει στις μεγάλες, στα έργα των, μεγαλών, ε, των υποδομών, στα μεγάλα έργα υποδομών. Ε, επίσης, η συμμετοχή, εμπλοκή των παραγόντων της κάθε περιοχής όταν πρόκειται να αναπτυχθεί ένα μεγάλο έργο ε, έργα όπως το κάστρο στην Ισπανία, γενικά της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, οι άλλες μεγάλες υποδομές, αυτοκινητόδρομοι, ε, σιδηρόδρομοι που περνούν από διάφορες περιοχές πρέπει να αναπτύσσονται σε συνεργασία και σύμπραξη με τους ε, πληθυσμούς αυτούς. Φανταστείτε δίπλα το σπίτι σα να αποφασιστεί να περάσει ένα αγωγό φυσικού αερίου. Προφανώς θα έχετε κάποιε αντιδράσει και ανησυχίε ενδεχομένω. Γι' αυτό πρέπει και οι κάτοικοι των περιοχών να συμμετέχουν στην προετοιμασία αυτών των σχεδιασμών για τα μεγάλα έργα που μπορεί να είναι και ε, επικίνδυνα ή πάντως όχι χρήσιμα για τους πληθυσμούς των περιοχών μας από τις οποίες περνούν και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται. Για τον ε, μοναδικό μειοδότη, single bidder, Οπωσδήποτε χρειάζεται καλύτερη πρόσβαση στα δεδομένα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες ως προς τον εντοπισμό των στοιχείων που έχουν να κάνουν με, ε, την, ε, με τις πρωτοβουλίες αυτές Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κάποια άλλα στοιχεία. Έξω θα ήταν καλό η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μελλοντικέ συναντήσεις να πρέπει να κληθεί για να μας δώσει, να μας επιβεβαιώσει τα στοιχεία. Και υπόθηκε ήδη ότι πρέπει να βελτιωθεί και το σύστημα της ε, πρόσβασης από πλευράς του πολίτη το σύστημα που επιτρέπει την πρόσβαση του πολίτη στις βάσεις αυτές, αυτά τα 20 δισεκατομμύρια που οι πολίτες διαθέτουν για την εκτέλεση των ε, μεγάλων έργων υποδομών, για τις ε, προμήθειες των δημοσίων αρχών των κρατών μελών, πρέπει να αξιοποιούνται σωστά. Ε, Κλείνοντα, θα ήθελα να πω ότι πρέπει και τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα τη αξιολόγηση, τη διαχείριση των μεγάλων αυτών έργων υποδομών. Πρέπει να τα στηρίξουμε λοιπόν ώστε να καλύψουν και τα σχετικά κενά. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσφέρει πληροφορίε, να προσφέρει δυνατότητε συνεργασία, ώστε να αναπτυχθούν οι βέλτιστε πρακτικέ σε επίπεδο κρατών μελών και ε, οπωσδήποτε και η διαφάνεια στη διαδικασία της προκήρυξης του έργου. Άρα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ κράτου κράτους-μέλους, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συντάκτες ε, της μελέτης. Βλέπω ότι η πρόεδρος ε, Γκρέσλε έχει ήδη εντοπίσει κάποια σημεία ε, επίκριση, αν και οι άλλοι συνάδελφοι έχουν κάποιε παρατηρήσει. Πολύ ευχαρίστω να τι ακούσουν, να τι λάβουμε υπόψη, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να κάνουμε εξαιρετική δουλειά πάντα στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Ευχαριστώ. Βεβαίως, βεβαίως και ευχαριστώ πολύ οι συνάδελφοι, θέλουν το λόγο. Αν όχι, θα παρακαλέσω τους δύο ε, εμπειρογνώμονες, τους δύο συντάκτες της έκθεσης να λάβουν το λόγο. Έχετε ιδιαίτερα εστιαστεί στα μεγάλα έργα, πάνω από 50 εκατομμύρια. Οπωσδήποτε η εικόνα θα είναι διαφορετική από αυτήν των μικρότερων έργων, γιατί 50 εκατομμύρια δεν μπορεί να τα ε, καλύψει κάθε επιχείρηση οπωσδήποτε ενδέχεται να είναι πάντα οι ίδιες επιχειρήσεις αυτές οι οποίες είναι σε θέση να αναπτύξουν τέτοια μεγάλα έργα. Παρακαλώ λοιπόν ε, να απαντήσετε για να ακούσουμε και, για τα, και από το κομμάτι που αφορά τα περιφερειακά. Ευχαριστώ πολύ για το θέμα της διαφοράς των δεδομένων και αναφέρθηκε νομίζω σε έναν βαθμό στην έκθεσή μας. Ένα στοιχείο λοιπόν είναι ότι έχουμε στηριχθεί στα ε, δεδομένα που κατεβάσαμε από το TNT και ενδέχεται τα εθνικά συστήματα ε, προκηρύξεων να έχουν πιο ακριβή στοιχεία. Από εκεί μπορεί να προκύπτουν ε, οι διαφορές, Γιατί η ανάλυση στην οποία προβαίνει η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακών Υποθέσεων δεν ξέρω τι στηρίζεται. αλλά δεν θα με εξέπλητα αν υπήρχαν διαφορές σε σχέση με ε, την, ε, τις βάσεις δεδομένων των κρατών μελών για τις προκηρύξεις τους, γιατί το τεστ είναι ένα είδος αναγγελίας, μια πλατφόρμα αναγγελιών. Ενώ τα εθνικά συστήματα, ελπίζουμε τουλάχιστον, έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να καταγράφουν στην πληρότητά τους, τις ίδιες τις συμβάσεις, ε, τις εκτελέσεις των ποσών κτλ. Και ακόμη, να συμπληρώσω, λέει ο κύριος Παπή, ότι έχουμε δει ένα 42% να λείπει σε σχέση με τις αξίες που καταγράφονται. Άρα τα σύνολα στα οποία εμείς ε, έχουμε καταλήξει έχουν τα ε, ποιοτικά τους όρια. Και πρέπει να τα δεχθούμε όπως έχουν. Στην σελίδα 51 της μελέτης, αν μου επιτρέπετε να σας ε, επιστήσω την προσοχή, στη μελέτη μας θα δείτε και την ανάλυση που αναφέρεται στο ιδιαίτερο, ε, στα στοιχεία τα συγκεκριμένα που λείπουν από τις μελέτες αυτές. Ναι. Και κάτι ακόμη. Κοιτάξτε, κάτι που δεν ανέφερα πριν. Στο TED έχουμε τριών ειδών συμβάσεις που ανατίθεται εφοδιασμό, υπηρεσίες και έργα. Ο εφοδιασμός ήταν πολύ ψηλότερος όσον αφορά τις ε, αναθέσεις αυτές με μοναδικό μειοδότη και ήταν μικρότερο ποσοστό της ε, ομάδας αυτών των συμβάσεων. Ευχαριστώ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριο Δένης από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακών Θεμάτων, παρακαλώ. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα ευχαριστώ και τους συμβούλους, να ευχαριστήσω τους συμβούλους για την πολύ καλή αυτή έκθεση. Ακούσα μεγάλο προβληματισμό της συλλογής στοιχείων. Στην καθημερινή μας δουλειά, αξιολογώντας τα έργα, έχουμε παρόμοια προβλήματα με στοιχεία που δεν συμπληρώνονται σε άλλα συστήματα, δεν εισάγονται. Και καθημερινά πολεμάμε για να βελτιώσουμε την εισαγωγή στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές των δικαιούχων κρατών μελών. Έτσι μπορούμε να προβούμε σε μια καλύτερη ανάλυση. Τώρα στις συστάσεις θα ήθελα να αναφερθώ σε λίγο. Πριν από αυτό να επενθυμίσω κάτι στην Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καταβάλουν προσπάθειες όσον αφορά την προετοιμασία των έργων. Έχουμε την πρωτοβουλία Jaspers, 140 άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αξιολογούν, παρέχουν συμβουλές για την προετοιμασία των έργων και τα αξιολογούν εν συγκρίση με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις και στην πολιτική συνοχής και με το μέσο για τη διασυνστημότητα της Ευρώπης, Connecting Europe Facility. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε την προετοιμασία ε, των έργων. Ε, δεν είναι τέλεια διαδικασία, χρειάζεται δουλειά ακόμα. Όπως αναφέρθηκε μετά, στη διαφάνεια που είδαμε, Είχαμε σχέδιο δράσης για τις κρατικές προμήθειες. Πολλές γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετείχαν. Δώσαμε πολλές πληροφορίες. Τις ε, δώσαμε στα κράτη-μέλη. Απογοητεύομαι κάπως διότι οι σύμβουλοι διαπίστωσαν τα κράτη-μέλη δεν ζητούν πληροφορίες, δεν τις χρησιμοποιούν όταν τις έχουν. Ίσως πρέπει να δούμε πώς θα μπορούσαμε να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να ωφεληθούν περισσότερο από αυτά που έχουμε κάνει και τις προσπάθειες που καταβάλουμε. Όσον αφορά τις συστάσεις, για την πρώτη σύσταση έχω να πω κάτι. αναφέρει ουσιαστικά στο σχέδιο δράσης για τις κρατικέ προμήθειες. Κάνουμε μελέτες πάνω σε αυτό. Καθημερινά αξιολογούμε τα μεγάλα έργα υποδομών. Συλλέγουμε στοιχεία συνεχώς. Εξετάζουμε τα έργα που εκτελούνται για να δούμε πόσο καλή προετοιμασία έχει γίνει. Όσον αφορά για τις επιδόσεις των διαφόρων πρωτοβουλειών και τα στοιχεία που συλλέγουμε από αυτών, δεν ξέρω αν τώρα είναι η στιγμή να ασχοληθούμε με αυτό. Είναι πρόσφατα τα στοιχεία και χρειαζόμαστε μεγαλύτερη εμπειρία. Όμως, μπορούμε να λάβουμε υπόψη τη σύσταση τη σχετική. Δυσκολότερο είναι το πρόβλημα της ασυνέπειας των στοιχείων του TED. Συμπληρώνται τα στοιχεία από την συμβαλόμενη αρχή. δοθέντος του αριθμού των στοιχείων που εισάγονται στη βάση δεδομένων, TED, δεν νομίζω ότι κάποιο ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο μπορεί να διεξαγάγει ποιοτικό έλεγχο επί των πληροφοριών. Όπως λένε και και ειδικοί ε, για την πληροφορική, άμα βάλεις σκουπίδια στο σύστημα, σκουπίδια θα βγάλει το σύστημα. Μπορεί να ζητήσουμε τα κράτη-μέλη να προσπαθήσουν, αλλά τελικά οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους καλύτερα. Τέλος. Πρέπει να πω ότι στην αρχή της παρουσιάσεως αναφερθήκατε στους διαφόρους ρόλους των διαφόρων εμπλεκομένων φορέων. Είπατε ότι πρέπει να ενισχυθεί η συμμετοχή των ενδιαφερομένων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να τους ενθαρρύνει, αλλά μόνο σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να δρομολογηθεί αυτή η δράση. Έτσι θα εξασφαλίσουμε ότι θα συμμετέχουν περισσότερο εμπλεκόμενοι φορείς. Το ρυθμιστικό πλαίσιο χρειάζεται ενίσχυση. Όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμμορφώνονται με την οδηγία για τις κρατικές ε, προμήθειες και οι συνάδελφοι στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης ασχολούνται με αυτό, κατά πόσο υπάρχει συμμόρφωση με την αρμόδια ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν ξέρω πόσο καλά μπορούμε να εντάξουμε σε αυτή την προσπάθεια το ρυθμιστικό πλαίσιο. Τροφή προσκέψη η μελέτη, χρησιμότατη. Λυπούμε που έχετε προβλήματα με τη συλλογή των στοιχείων και είδαμε κάποια στοιχεία που είναι σαφώς γελία παρά τους περιορισμούς που δημιουργούνται από τα στοιχεία και τα δεδομένα είναι χρήσιμη η μελέτη και θα τη λάβουμε υπόψη και θα τη μελετήσουμε συνεχίζοντας τις προσπάθειές μας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα και κυρίως δεν κατάλαβα για ποιο λόγο η μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης περιφερειακής ανάπτυξης για το ίδιο θέμα αφίσταται τόσο πολύ από τη σημερινή μελέτη και έχουν τέτοιες διαφορές στα αριθμητικά στοιχεία και δεν μας είπατε τίποτα. Και επίσης δεν κατάλαβα γιατί δεν είναι καλύτερη η κατάσταση των δεδομένων και ποιος φταίει. Δεν έχουμε ε, επαρκή στοιχεία, είμαστε τόσο ανίκανοι που δεν μπορούμε να τα συλλέξουμε. Τα δεδομένα. Πού είναι το πρόβλημα. Αν θέλετε ξαναπείτε τα από την αρχή γιατί εγώ δεν κατάλαβα καθόλου. Ε, και δεν με ικανοποιεί η σημερινή συζήτηση επίσης καθόλου. Βλέπουμε τεράστια ποσά να διακινούνται και η επιτυχία ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εσωτερική ε, αγορά είναι η διαφάνεια των διαδικασιών. Πού είναι εδώ η διαφάνεια των διαδικασιών. Είναι σκέτο χάλι κατάσταση με τα δεδομένα. Παρακαλώ, έχετε ξανά το λόγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας το εξηγήσετε. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να σας διαφωτίσω. Αν θα τα καταφέρει όχι, δεν γνωρίζω. Τι μπορούμε να κάνουμε. Μόλις λάβαμε την έκθεση βλέπετε. Άρα πρέπει να συγκρίνουμε την έκθεση με τα στοιχεία που περιέχει και να τα συγκρίνουμε με τα στοιχεία που έχουμε στην, στην Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης και να δούμε γιατί υπάρχει αυτή η απόκληση στοιχείων, που είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σήμερα δεν μπορώ να δώσω απάντηση. Μπορούμε να κάνουμε κάποια ανάλυση για να δούμε γιατί υπάρχει διαφορά στα αποτελέσματα και να δούμε αν μπορούμε να εντοπίσουμε που υπάρχει το πρόβλημα με τα δεδομένα. Εάν έχουμε ερωτήσεις από αυτά που παρουσίασαν οι σύμβουλοι στις διαφάνειες, θα απευθυνθούμε σε αυτούς. Θα το ψάξουμε με άλλα λόγια να δούμε γιατί υπάρχει αυτή η μεγάλη απόκληση μεταξύ των δεδομένων. Ευχαριστώ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Για μια στιγμή. Έχουμε τη μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακών Υποθέσεων. Προσωπικά την έχω αξιολογήσει και λέγει αυτή η μελέτη ξεκάθαρα ότι ε, υπάρχουν διάφορα στάδια ε, στην προκήρυξη του διαγωνισμού και καταλήγει σε διαφορετικά συμπεράσματα για την Ουγγαρία, για την Πολωνία, γιατί απορροφούν πολλά κονδύλια. Γι' αυτό θα ήθελα να το εξηγήσετε. Πόθεν ε, τα διαφορετικά αριθμητικά στοιχεία και πού είναι το πρόβλημα. Εγώ δεν ασχολούμαι για την πλάκα μου με αυτά τα θέματα. Ε, θέλω και ε, απαντήσεις. Το ωραίο και το καλό είναι ότι τα διαβάζουμε όλα αυτά που μας στέλνετε. Τα διαβάζουμε και τα συζητάμε εδώ και μήνες και προσπαθούμε να κατανοήσουμε για ποιο λόγο σε κάποια κράτη-μέλη στις μισές ε, διαδικασίες και τα έργα. Δεν υπάρχει δεύτερος ε, υποψήφιο στην προσφορά μειοδότης και αυτό ονομάζεται διαφθορά, έχει όνομα. Να τα λύσουμε, να δούμε που θα καταλήξουμε τα στοιχεία. Πραγματικά πρέπει να σας πω ότι με έχετε κατά Αν θέλετε πάρτε και πάλι το λόγο, αλλά θέλω να μου πείτε κάποια πράγματα περισσότερα. Παρακαλώ. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως σας είπα, μόλις λάβαμε την έκθεση. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε τις κατάλληλες συγκρίσεις με πρώτερες δικές μας μελέτες. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Σήμερα δεν μπορώ να δώσω απάντηση και εξήγηση. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά στα αποτελέσματα γιατί τα ποσοστά με μοναδικό μειοδότη διαφέρουν τόσο πολύ. Δεν μπορώ σήμερα να σας δώσω απάντηση. Λυπάμαι πάρα πολύ. Είναι θέμα να κάνουμε σωστή δουλειά. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Χρειάζεται διαφάνεια. Θα πρέπει να έχουμε δεδομένα που να είναι σωστά. Για να έχουμε σωστά αποτελέσματα. και για να μπορούμε να κατανοήσουμε το τι συμβαίνει επί τόπου. Σήμερα όμως δεν μπορώ να εξηγήσω αυτές τις διαφορές. Λυπούμε. Πρέπει να εξετάσουμε τη μελέτη και να τη συγκρίνουμε με τη δική μας, αυτή που κάναμε. Και πότε με το καλό να σας ξανακαλέσουμε, πότε θα είστε έτοιμοι. Um, Κοιτάξτε, θα χρειαστούμε κάποιες εβδομάδες, δύο-τρεις μήνες. Αρχές του επομένου έτους, το πρώτο τρίμηνο του επομένου έτους μπορούμε να προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποια απάντηση. Με χαρά να τα ξαναπώ με το Μάρτιο, θα το γράψουμε και πάλι στην ημερησία διάταξη, αλλά θέλω να μάθω από εσά, ε, από την εμπειρία σας, γιατί πόσο καιρό εργάζεστε σε αυτό το κλάδο κατά την εμπειρία σας. Επαρκεί το κανονιστικό και το ρυθμιστικό πλαίσιο. Είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν ε, αυτές τις διαδικασίες. Είναι επαρκής αυτή η διαδικασία. Προβλέπετε και στο νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο ή σας είναι όλα διάφορα. I think we have... Κοιτάξτε. Έχουμε αντικρουόμενες δυνάμεις εδώ. Τις δυνάμεις που θέλουν πλήρη διαφάνεια, που συνεπάγεται πολλές πληροφορίες. Πολλές πληροφορίες συνεπάγονται περιπλοκές, βάρος, τις αρμόδιες αρχές, δικαιούχους, κράτη, μέλη, χρειάζονται ε, δυνάμεις και πόροι και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αλλού. Από την άλλη πλευρά έχουμε τη δύναμη της απλούστευσης, όπου οι κανόνες είναι απλούστεροι και αν οι κανόνες είναι απλούστεροι, θεωρητικά είναι ευκολότερο να συμμορφωθεί κανείς. Εθελοντικά υποβάλλονται οι πληροφορίες. Δεν υπάρχει μια νομική βάση ξεκάθαρη και αυστηρή για να υποβάλλονται οι πληροφορίες και ενημέρωση μέσω πυθούς και μέσω διαφόρων τεχνικών, συναντριάσεων εμπειρογνωμόνων, μέσω μελετών μπορούμε να συλλέξουμε τις αναγκαίες πληροφορίες. Από μία πρώτη ματιά πρέπει να πω ότι δεν χρειάζεται να επιβληθούν συμπληρωματικέ υποχρεώσεις υποβολής πληροφοριών από τα κράτη-μέλη ή από τις αρμόδιες αρχές σε αυτό το στάδιο. Άρα μπορούμε να μάθουμε περισσότερα, αν το θέλουμε, αλλά μου φαίνεται ότι δεν θέλουμε να μάθουμε περισσότερα. Ε, πολύ δυσάρεστη εντύπωση που μου προξενεί, γιατί ξέρουμε ότι είναι πολλά τα κονδύλια που έχουν προβλήματα, όχι μόνο λόγω διαφθοράς ή αδιαφάνειας, αλλά και γιατί υπάρχει αυτή η αδιαφανειας αλλα και γιατι υπαρχει αυτη αδυναμία να αξιοποιηθούν σωστά και αυτό το οποίο είπε και ο κύριος Βάλη δυστυχώς θα πρέπει να το επαναλάβω ότι με την διαφάνεια μπορούμε να δώσουμε απάντηση στις κατηγορίες που απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μου κάνει καθόλου καλή εντύπωση όλη αυτή η ιστορία. Το Μάρτιο τα ξαναλέμε, δεν σας ξεχνώ. Και ερωτώ τους ε, στάκτες έκθεση αν θέλουν να προσθέσουν κάτι ακόμη. Ευχαριστώ πολύ. Και το σημαντικό πιστεύω εδώ είναι το τι δεδομένα ε, έχει χρησιμοποιήσει για ως βάση ανάλυσης αλλά και τη μεθοδολογία η Γενική Διευθυνσία Περιφερειακών Υποθέσεων. Εμείς, σε παραδείγμα, τα δεδομένα ΤΕΚ δεν μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να αντλήσουμε στοιχεία για συγκεκριμένα κονδύλια. Απλώς μας ε, δίνει μια ένδειξη αν υπήρξε ανάμειξη και ευρωπαϊκών κονδυλίων ή όχι σε ένα συγκεκριμένο έργο. Άρα λοιπόν θα πρέπει ίσως να συγκρίνουμε τις μεθοδολογίες μας και τις πηγές των δεδομένων ε, για να εντοπίσουμε αν κοιτάμε, μελετούμε το ίδιο σύνολο συμβάσεων. Γιατί σε αυτό το στάδιο που είμαστε δεν μπορούμε να γνωρίσουμε αν, να γνωρίζουμε αν πρόκειται για τις ίδιες πληροφορίες, αν η μελέτη μας στηρίζεται στο ίδιο σύνολο πληροφοριών. Μπορεί να έχουμε και διαφορές στις μεθοδολογίες. Επομένω θα ήταν καλό να μπορούμε να κοιτάξουμε αυτό. Η πρόεδρος, ε, ναι, εντάξει, αλλά ένα λεπτό, το αντικείμενο είναι το ίδιο. Πόσε επιχειρήσει έχουν λάβει μέρο σε έναν ευρωπαϊκό ε, διαγωνισμό. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι πληροφορίες και με βάση τις ε, και οι μελέτε δηλαδή τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακών, αλλά και οι δικοί σα πρέπει να έχουν αντίστοιχα. Δεν μπορεί να έχουν τόσο διαφορετικά αποτελέσματα. Γι' αυτό λοιπόν και σε μεγάλη αμηχανία ε, και απορία βρισκόμαστε. Και θεωρούμε ότι κάπου πρέπει να υπάρχει ένα σφάλμα. Δεν είναι δυνατόν με το ίδιο αντικείμενο μελέτης να έχουμε τόσο μεγάλη διαφορά στα αποτελέσματα. Τουλάχιστον δική μου εμπειρία αυτό λέει. Αυτό λοιπόν. Θέλω πιο σαφείς απαντήσεις και δίνω το λόγο, αν δεν θέλετε κάτι να προσθέσετε, στον εισηγητή. Κύριος Βάλη. Ναι, πάντως, Μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένο ε, που επισημάνθη πως θα γίνουν περαιτέρω ε, παληθεύσεις και ε, μελέτες ως προς τα αποτελέσματα των εργασιών. Προσπαθήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκαθαρίσει ορισμένα πράγματα. Έργα μεγάλα, δεν θα τα πω και φαρανοϊκά, φαραωνικά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σημαντικά πολύ μεγάλα έργα, μπορεί να κρατούν χρόνια και είναι απαραίτητο να ξέρουμε ότι με ό,τι αλλαγές μπορεί να έχουν υπησέλθει σε επίπεδο ονομάτων ή προσωπικότητων νομικών των επιχειρήσεων, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα διαφάνειας κτλ. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει δυνατότητα να μας δίνουν και η Επιτροπή και οι υπεύθυνοι των μελετών, όποιες είναι αυτές, στοιχεία σαφή, χωρίς τα προβλήματα αυτών των διαφορών που εντοπίσαμε. Είναι σημαντικό να το συζητούμε λοιπόν. Χωρίς διάλογο, χωρίς συζήτηση, τα λάθη θα επαναλαμβάνονται. Όταν εντοπίζουμε λοιπόν τα, τις δυσκολίες, ελπίζουμε ότι μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και γι' αυτό ευχαριστώ και την Πρόεδρο που πάντα επιμένει για τις λεπτομέρειες που εντοπίζει στα προβλήματα τα σχετικά με τα δεδομένα στα οποία συζητούμε στηρίζονται οι μελέτες και βεβαίως τον Μάρτιο θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε. Σας ευχαριστώ και εσάς, η Πρόεδρος. Εντάξει, το κρατάμε ανοιχτό το θέμα. Το αφήνουμε για το Μάρτιο. Και περιμένουμε σαφείς απαντήσεις για το σημαντικό αυτό θέμα. Σημαντικό για μας, σημαντικό γενικώ και γιατί έχει να κάνει και με την απρόσκοπτη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στο θέμα των ε, διαγωνισμών των δημοσίων προμηθειών. Αυτά. Κλείνει εδώ το θέμα αυτό τη ημερήσια διάταξη. Δεν ξέρω αν ο Γενικό ε, Γραμματέα μας περιμένει, είναι αντεπόρτας ή αλλιώ να διακόψω μέχρι την άφηξή του. Συνεχίζουμε με την ημερήσια διάταξη. Απαλλαγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καλωσορίζω τον συνάδελφο σα όλοι, αντιπρόεδρο αρμόδιο για τον Προπολογισμό και τον Γενικό Γραμματέα Βέλα, τον εσωτερικό ελεγκτή, τον κύριο Γκάλβιν και εκπροσωπεί τον κύριο Ρούσο που ασθενεί και ε, ε, ε, έχει έρθει η κυρία Τσιπριάνη, διευθύντρια του ε, γραφείου του και θα μας παρουσιάσει αμέσως το αντίστοιχο κεφάλαιο ε, της έκθεσης ε, του ελεγκτικού συνεδρίου. Προηγουμένως όμως και στα γαλλικά θα ήθελα να καλωσορίσω ομάδα επισκεπτών από τον Νίγηρα και την ακτή Ελεφαντοστού. Είναι συνάδελφοι από τη Βουλή των δύο χωρών, της κάστοτε χώρας. Καλωσορίσατε. Χαιρόμαστε ε, που σας έχουμε ενώπιον μας και ελπίζω να βρείτε ενδιαφέροντα τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα θέματα αυτά της απαλλαγής και της λογοδοσίας. Το λόγο έχει η κυρία Τσιπριάνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και άρα Τσιπριάνη. Λέγομαι και είμαι. Με ακούτε έτσι. Επικεφαλής του ε, επιτέλειο του κύριου Ρούσο. Στο συγγνώμη που δεν μπόρεσε να παραστεί σήμερα στη συνεδρίαση και την ακροασή σας για λόγους υγείας. Θα κάνω την παρουσίαση λοιπόν του κεφαλαίου υπαριθμών 10 της ετησίας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και την αξιολόγηση των διοικητικών δαπανών, ιδιαίτερο σήμερα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η έκθεση λοιπόν καταλήγει σε θετική αξιολόγηση. Οι δαπάνες δεν σημειώνουν σημαντικό ε, ποσοστό σφάλματος. Το εκτιμούμενο ποσοστό είναι 0,5%. Αυτή η αξιολόγηση στηρίζεται σε δείγμα 55 μεταφορών κονδυλίων, εκ των οποίων οι 11 έχουν να κάνουν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τέσσερις εκ των συναλλαγών ή πληρωμών βλέπουμε να παρουσιάζουν σφάλμα. Συνολικά έχουμε επτά σφάλματα διαφορών ειδών, μεταξύ των οποίων έχουμε ποσοστικά μετρήσιμο σφάλμα στην καταβολή μη επιλέξιμων δαπανών για ομάδα επισκεπτών. Οι άλλε έξι κατηγορίε σφαλμάτων έχουν να κάνουν με αδυναμίες ω προς τον εντοπισμό των διαδικασιών ε, δημοσίων προμηθειών, το μη σεβασμό του χαρακτήρα του ενιαύσιου, του προπολογισμού, αλλά και ανεπαρκής εκ των προτέρων ελέγχων, αλλά, ελέγχους, αλλά και εκ των υστέρων ανεπάρκειες στις επαληθεύσεις ε, των ε, τιμολογίων των δαπανών. Και έτσι λοιπόν ε, συγκεκριμένα συνιστούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βελτιώσει τις κατευθύνες γραμμές για την χορήγηση για τους ε, ε, διατάκτες ως προς το σχεδιασμό και τις επαληθεύσεις των κριτηρίων επιλογής και χορήγησης των διαδικασιών των προμηθειών. Επίσης, συνιστούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν πρόκειται να αναθεωρήσει τους κανόνες που διέπουν την υποδοχή ομάδων επισκεπτών να ενισχύσει τη διαδικασία για την υποβολή δηλώσεων δαπανών, απαιτώντας από τις ομάδες να, ε, των επισκεπτών να καταθέτουν τα σχετικά αποδεικτικά μαζί με τις αιτήσει για επιστροφή εξόδων. Επίσης έχουμε αξιολογήσει την ε, συνέχεια που δόθηκε στις γενικές συστάσεις ε, που είχαμε διατυπώσει με την ετήσια έκθεση του 2014. Ε, σε σχέση με τους μισθούς και, τις, και τα οικογενειακά επιδόματα βλέπουμε ότι οι συστάσεις μας έχουν γίνει σεβαστές επιτοπλίστων σε σχέση με τη σύσταση που έχει να κάνει με την ενίσχυση των ελέγχων για την επιστροφή δαπανών και το σεβασμό των ε, αρχών και κανόνων για τη διεξαγωγή δημοσίων ε, προκηρύξεων από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί ε, δυνατότητα για ανάλυση, δική ανάλυση της πρόοδου που έχει πραγματοποιηθεί. Κυρία Πρόεδρε, μας θέσή σας για περαιτέρω διευκρινή. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αρχίζουμε τον κύριο Σασόλη, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και απαντήσατε και σε ένα ερωτηματολόγιο, κύριε Γενική, με 161 ερωτήσεις. Κύριε Σασόλη Σασόλ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι. Λοιπόν, είμαστε στην απαλλαγή για τον προπολογισμό 2017 και θέμα στο δυνατόν λακωνικός και θα ομαδοποιήσω τις ερωτήσεις μου σε διάφορα θέματα για να εξασφαλίσουμε στο δυνατόν περισσότερες πληροφορίες βεβαίως. Το 1,91 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ για τον προϋπολογισμό του 2007 έχει κατά 99% απορροφηθεί και ε, ένα 0,1% μόνο φαίνεται να έχει πρόβλημα. Ε, άρα νομίζω ότι έχουμε πολύ καλές επιδόσεις να καταγράψουμε σχέση και με τις ε, προβλέψεις για τον προπολογισμό και την εκτέλεση από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο οφείλουμε και στην προκαταβολή ποσών και τη μεταφορά 40,85 εκατομμυρίων από το έργο του ΚΑΔ κτηρίου στο Λουξεμβούργο με την άδεια που χορηγήθηκε από την Επιτροπή των Προϋπολογισμών και που μας επέτρεψε έτσι να εξοικονομήσουμε ε, από τόκους 8,3 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ αυτό. Για την ασφάλεια. Το έργο για την ενίσχυση της εξωτερικής ασφάλειας των κτηρίων μας ξέρω ότι ξεκίνησε το 2017 ιδιαίτερα σε συνεργασία και με τις εθνικές αρχές που μας φιλοξενούν μπορέσαμε να δημιουργήσουμε ε, περιφέρειες ασφαλείας γύρω από τα κεντρικά μας κτίρια, ιδιαίτερα στις Βρυξέλλες. Έχουμε την πεζοδρόμηση της οδού Βίρτσα, ε, καθώς αποτελούσε σημαντικό κίνδυνο, ε, παράγοντα κινδύνου η κυκλοφορία των οχημάτων. Επίσης ενισχύεται η ασφάλεια στις εισόδους ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με βάση και τα όσα είχαν αποφασιστεί το 2016 και πραγματοποιηθεί στο κτίριο Σπινέλη ήδη. Ε, με τον περιορισμό λοιπόν και του παράγοντα κινδύνου για τους βουλευτές και το στόχο αυτό αποφασίστηκε η ε, εσωτερική οργάνωση μιας υπηρεσίας ε, οδηγών με καλύτερη δυνατότητα έλεγχου ως του προσωπικού αλλά και τη δυνατότητα στους εργαζόμενους μας να προσφέρουμε κατάλληλες συνθήκες εργασίας. 116 ήταν αυτοί οι οποίοι προσλήφθηκαν με δημόσια προκήρυξη των θέσεων. Ε, κτίρια τώρα στο ΚΑΝΤ του Λουξεμβούργου συνεχίζονται οι εργασίες χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Κάποιες αναφορές ε, πρόσφατες μας ε, δίνουν δαπάνες κάτω των 38,32 εκατομμύριων που είχαν αρχικά προβλεφθεί. Στο Στρασβούργο το, το άνοιγμα του, και η χρήση του κτηρίου Παύελ, θα μας δώσει περισσότερους χώρους στη διάθεσή μας και άρα περισσότερο περιθώριο για ε, διάθεση γραφείων στους βουλευτές. Απαραίτητε οι χώροι βεβαίως όλοι αυτοί για να γίνεται καλά η δουλειά των βουλευτών, καθώς πολύ συχνά στο Στρασβούργο υποχρεούνταν οι ευρωβουλευτές να μοιράζονται το γραφείο τους μαζί με τους βοηθούς του ή άλλο προσωπικό, πράγμα το οποίο περιόριζε βέβαια και τις δυνατότητες ε, αποτελεσματικής δουλειάς, αλλά και τον ιδιωτικό τους χώρο και βίο. Στο Στρασβούργο το κτίριο Μάρτενς μας δίνει με την ε, θέση του σε Τουρκία επιτρέπει την απελευθέρωση πολλών χώρων και γραφείων. Πράγμα πολύ σημαντικό καθώς τα τελευταία χρόνια το προσωπικό μας έχει αυξηθεί. Έχουμε περισσότερους βοηθούς, ε, ασκουμένους, όλους αυτούς τους οποίους οφείλουμε να προσφέρουμε κατάλληλες συνθήκες εργασίας. Οι υβριδικοί υπολογιστές και η ε, χρήση νέων λύσεων, η δοκιμή δοκιμαστική χρήση. Έχει ξεκινήσει λοιπόν μια δοκιμαστική χρήση υβριδικών υπολογιστών από τη Γενική Διεύθυνση ΙΤΕΚ που έχει στεφθεί με εξαιρετική ε, επιτυχία και αποτελεί ε, μια νέα ιδέα κινητικότητας, υλοποίηση μιας νέας ιδέας κινητικότητας για να μπορούμε να έχουμε όλοι μας το γραφείο μας πάντα ε, αναχείρας. Τα γραφεία και ο εξοπλισμός των γραφείων, αλλά και ο νέος χώρος εργασίας για τους βουλευτές που θα έχετε ίσως δει σε ορισμένες αίθουσες του Κοινοβουλίου, ότι έχουμε αναπτύξει μικρές ε, αίθουσες ε, συνεδριάσεων με μεταξύ 8 και 10 ατόμων, όπου έχουν εγκατασταθεί τα απαραίτητα ώστε να φιλοξενεί ένας βουλευτής προσκεκλημένου του σε μικρή σύνθεση ε, συνεδριάσεις και εκεί έχουμε ακόμα και ε, μια μικρή ένα μικρό χώρο κουζίνας που μπορεί να αξιοποιηθεί και κρίνεται γενικά πολύ, θετικός, ε, από τους βουλευτές. Το υλικό, τα έπιπλα, που είναι αρκετά πεπαλαιωμένα και χρειάζονταν ανακαίνιση. Αντί λοιπόν να αγοράσουμε καινούργια, αποφασίσαμε την λύση της, ε, του, του leasing, ε, γιατί έτσι απαλλασσόμαστε και από την ε, υποχρέωση για επισκευές, ανακαίνιση κτλ. Και έτσι αυτή η λύση του leasing μας δίνει μια επιβάρυνση μηδενική για τον προπολογισμό, όχι ουδέτερο δηλαδή αποτέλεσμα αντίκτυπο στον προπολογισμό. Ε, στην ομάδα εργασίας και έχω δει και στο ερωτηματολόγιο κάποιες ερωτήσεις σχετικές με τα γενικά έξοδα των βουλευτών και φαντάζομαι ότι θα διατυπωθούν τα σχετικά ερωτήματα. Ε, καθώς είμαι πρόεδρος ε, της ομάδας εργασίας για την αναθεώρηση των κανόνων των σχετικών με την αποζημίωση γενικών εξόδων και δεδομένων και των ετοιμάτων που έχουν κατατεθεί, των προτάσεων μάλλον για την αναθεώρηση του προϋπολογισμού του 2018 που συγκεκριμένα αναφέρονταν στην ανάγκη να υπάρχει ένας χωριστός τραπεζικός λογαριασμός, επιστροφή των ε, ποσών που δεν έχουν δαπανηθεί και αποδεικτικά στοιχεία. Έχουμε, μια πρόταση, η οποία, έχουμε καταλήξει μια πρόταση που προβλέπει ένα μεικτό σύστημα, δηλαδή ένα ελάχιστο ποσό που θα δίνεται κάτω από κοπήν χωρίς αποδεικτικά και το μεγαλύτερο κομμάτι της γενικής αποζημίωσης θα ήταν με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία. Ξέρετε ότι αυτή είναι η πρότασή μου. Ξέρετε όμως ταυτόχρονα ότι έχασα αυτόν τον ε, αυτή την ε, μάχη και έτσι αναγκάστηκα και να παρετηθώ στην ομάδα εργασίας, από την ομάδα εργασίας ως πρόεδρος, ο πρόεδρος ο οποίος, ο συνάδελφος ο οποίος με αντικατέστησε έχει ακολουθήσει διαφορετική γραμμή. Η γραμμή η οποία ενεκρίθηκε, υποστηρίχθηκε από την πλειονότητα των ε, αντιπροέδρων ε, με βάση και τα όσα είχαν επιλέξει οι πολιτικές τους ομάδες. Ε, πιστεύω ότι το ψήφισμα του Κοινοβουλίου απαιτεί την εγκατάλειψη του καταποκοπήν συστήματος, ωστόσο το ψήφισμα αυτό δεν υποστηρίχθηκε από την πλειονότητα των βουλευτών και έτσι παρετήθηκα από πρόεδρος της ομάδας εργασίας. Σε σχέση με το ενοποιημένο ταμείο συντάξεων, συνταξιοδότησης. Πριν από 10 χρόνια περίπου είχε λάβει απόφαση το Προεδρείο όπου οριζόταν πως το Κοινοβούλιο θα αναλάμβανε την ευθύνη να αντικαταστήσει στις πληρωμές, να υποκατασταθεί μάλλον στις πληρωμές σε σχέση με το Σταξιδοτικό Ταμείο Άπαξ και αυτό δεν θα ήταν σε θέση να εκτελέσει υποχρεώσεις του μόνο του αν δεν λάβει νέους σπόρους. Δηλαδή γύρω στο 2024 θα εξαντληθεί ε, κάθε περιθώριο πληρωμής από πλευρά αυτού του Ταμείου και άρα θα πρέπει στον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προβλεφθούν οι πόροι εκείνοι που θα επιτρέψουν την αντιμετώπιση των πόρων που έχουμε, των δαπανών που έχουμε ήδη εγκρίνει. Αναζητήθηκαν διαφορετικές λύσεις σε επίπεδο ε, προεδρείου, λύσεις νόμιμες, νομότυπες που δεν θα μας οδηγούσαν από το Ευρωπαϊκό Δικαστηρίο και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καλύψει τις σχετικές δαπάνες. Για τους ε, βοηθούς των, ε, βουλευτών, των ε, έχουμε λοιπόν κληθεί να συζητήσουμε και να λύσουμε το πρόβλημα των πιστοποιημένων βουλευτών που παρότι έχουν επί δύο συνεχόμενες βουλευτικές θητείες ε, απασχοληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συμπλήρωναν 10 χρόνια που απαιτούνται για τις ε, ε, για την εξασφάλιση των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις ήδη που έχουν κατευθεί και θα τις αξιολογήσουμε για να καταλήξουμε σε μια θετική λύση. Όσον αφορά τον κανονισμό των ασκουμένων, θα ήθελα να τονίσω ότι και αυτό το θέμα μας απασχολεί, το επεξεργαζόμαστε κατά γενικό κανόνα θα πρέπει οι ασκούμενοι να ε, εργάζονται με αμοιβή. Πρέπει να προσδιοριστούν όρια χρονικά συγκεκριμένα για την διάρκεια των ε, πρακτικών ασκήσεων και η σύμβαση αυτή δεν θα πρέπει να μετατρέπεται σε μια ατυπική μορφή ε, εργασίας ή σύμβασης εργασίας που θα αντικαθιστά ουσιαστικά τη σύμβαση του διεπιστευμένου βοηθού. Αυτά και σταματώ εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γενικός Γραμματέας, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι ο αρμόδιος αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου τα παρουσίασε πάρα πολύ εμπεριστατωμένα και εξαντλητικά, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω εγώ. Μία ε, παρατήρηση μόνο. Το 2017 ήταν και ένα έτος μαζικών περικοπών θέσεων. 136 θέσεις αφήσαμε, 60 ε, που ε, απορρέουν από το 5% των μειώσεων και 67% ε, από επιπλέον θέσεις που είχαν οι πολιτικές ομάδες. Αυτό επηρέασε σημαντικά τις εργασίες μας. Θέλω να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο και πάλι για τις παρατηρήσεις. 0,5% ε, ήταν το ποσοστό σφάλματος, το οποίο δεν αξιολογείται. ευχαριστώ πολύ οι περικοπές προσωπικού το 2017 και το Συμβούλιο παρεύει τη Συμφωνία Κύριων. Ο κύριος Γκάλβιν, ο ιστορικός ελεγκτής, έχει το λόγο για να μας παρουσιάσει την έκθεσή του. Παρακαλώ. Ε, Κυρία Πρόεδρε και μέλη της Επιτροπής, καταρχάς να σε ευχαριστήσω κυρία Πρόεδρε, για τη δυνατότητα που μου δίνετε να παρουσιάσω την ετήσια έκθεσή μου για το έτος 2017. Ο δημοσιονομικός κανονισμός απαιτεί στο ιστορικός ελεγκτής να υποβάλει στο θεσμικό όργανο ετήσια έκθεση που αναφέρει τον αριθμό και το είδος εσωτερικών ελέγχων που διενεργήθησαν, τις συστάσεις που έγιναν και τη δράση που ανελήφθη βάσει αυτών των συστάσεων. Αυτή η έκθεση, συνεπώς, αφορά τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του εσωτερικού ελεγκτού το 2017. Το τμήμα 2 της εκθέσεως περιγράφει την αποστολή της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, τη φύση και το όριο των δραστηριοτήτων, τα επαγγελματικά πρότυπα με τα οποία συμμορφούνται και πώς είναι οργανωμένοι. Υπενθυμίζει ότι η ανεξαρτησία του εσωτερικού ελεγκτικού φορέα και η διεξαγωγή των ελέγχων ε, αποτελούν αντικείμενο εγγυήσεω μέσω τη νομοθεσία Ευρωπαϊκή Ενώσεω και αναφέρονται στην χάρτα του εσωτερικού ελεγκτή. Εκεί που εντοπίζονται δυνατότητες ή ελλείψεις, κάνουμε συστάσεις υπό τη μορφή προτινομένων δράσεων. Μέσω διαδικασίας συνεχούς διαλόγου και επικοδομητικής διαβουλεύσεως με την υπηρεσία που ελέγχεται, επιδιώκει να πετύχει συμφωνία με τη διοίκηση επί της ουσίας και του χρονισμού των εν λόγω δράσεων. Στο τρίτο τμήμα περιγράφεται το έργο το ελεγκτικό που έγινε το 2017 και εξηγεί ότι ο εσωτερικός ελεγκτής Κάθε ετήσιο πρόγραμμα το συντάσσει βάσει συστηματική αξιολογήσεω του κινδύνου όσον αφορά όλον τον οργανισμό. Βασικό σκοπό αυτή τη αξιολογήσεω του κινδύνου να δώσει δυνατότητα στο φορέα εσωτερικού ελέγχου να θέσει προτεραιότητε αφορά την κατανομή των πόρων προ του τομεί εκείνου που αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερο κίνδυνο και χρήζουν μεγίστη προσοχή. Θα ήθελα ακροθυγώ να περιγράψω τι διάφορε διάφορες, έργα που έγιναν το 2017. Ο έλεγχο τη Γενική Διευθύνσεω επικοινωνιών και οργάνωσης των προσκλήσεων για τους ε, δημοσιογράφους είναι ένα τμήμα ε, του φορέα ελέγχου στη στατηγική Πολιτού. ελέγχου. Αυτές οι προσκλήσεις στις συνόδους και σε εκδηλώσεις και στις Βρυξέλλες του Στρασβούργου έχουν σαν στόχο να προωθήσουν τη διάδοση των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου στα μέσα ενημέρωσης. Η ελεγκτική στόχη ήταν να αξιολογηθεί η συμμόρφωση της διαδικασίας για την οργάνωση των προσκλήσεων με το ρυθμιστικό πλαίσιο και να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της εν λόγω διαδικασίας. Παδεχόμενη την αφοσίωση τη Γενική Υψήσεω Επικοινωνία για την επίτευξη αυτών των στόχων, ο εσωτερικό έλεγχο βρήκε και πεδίο ε, βελτιώσεω διαχειρήσεω και του ελέγχου και του συντικού πλαισίου σε τέσσερι τομεί. Πρώτα απ' όλα, ενίσχυση του πλαισίου, τόσο ώστε να αυξηθεί η εξασφάλιση του ότι οι αποζημιώσει προς τους δημοσιογράφους ευθυγραμμίζονται με το πραγματικό κόστος που διαπιστώθηκε. Δεύτερον, οι συστημικές αποκλήσει από τους κανόνες που διέπουν τις προσκλήσει να καλυφθούν να βελτιωθεί αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα ε, των λογιστικών, των σχετικών καταβάλλοντα πληρωμές ε, υποχρεωτικά μέσω εμβασμάτων τραπεζικών, Κατευθυντήριε γραμμέ για να αποσκαλούνται οι δημοσιογράφοι, ούτως ώστε να υπάρχει καλύτερη διάδοση των πληροφοριών όσον αφορά τη διαδικασία αυτή που πρέπει να γίνει πιο οικονομική αποτελεσματική. Οπότε ο εσωτερικό έλεγχο συμφώνησε επ' ενό σχεδίου δράσεω ε, με τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνία ε, με 11 σημεία. Θέλουμε να καλυφθούν οι τομεί μετρίου κινδύνου και σοβαρού κινδύνου. Τέσσερι δράσει για το σοβαρό κίνδυνο. Σαν ισοπρόθεσμη στρατηγική για τον έλεγχο όλων των σημαντικών διαδικασιών και των διαφόρων διευθύνσεων που ασχολούνται με την δαπάνη προσωπικού, ο εσωτερικό έλεγχο έκανε την το πρώτο έλεγχο από δύο ελέγχους για τα διάφορα ευεργετήματα, τα ατομικά, σύμφωνα με τον κανονισμό προσωπικού και τους κανονισμούς περί αυτό αφορά ε, τα ταξιδιωτική αποζημίωση, η καθημερινή αποζημίωση και τα αποζημίωση για εκπατρισμό. Στόχο είναι να αξιολογηθεί η συμμόρφωση για την ε, επίδοση των ευεργετημάτων αυτών σύμφωνα με του κανόνε και να γίνει η αξιολόγηση κατά πόσο τα συστήματα ελέγχου αποδοτικά. Ο εσωτερικό έλεγχο παραδέχεται ότι ήταν θετικά κάποια μέτρα που η Γενική Διεύθυνση Προσωπικού για να εξυγχρονιστεί η διαδικασία λήψη αποφάσεων επίση βρήκε ότι υπάρχει πεδίο για να καλυφθούν διάφορα προβλήματα στο κάτω θητομή. Χρειάζεται βελτίωση στο περιβάλλον του ελέγχου και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για του ελέγχου συμπεριλαμβανομένων σημαντικών προβλημάτων πρέπει να επιληθούν όσον αφορά την πληροφορική, κάτι που συνδέεται με το σύστημα διαχείριση του προσωπικού. Δεύτερον, χρειάζεται χρειάζονται ειδικέ διαδικασίε για το προσωπικό και διαχείριση όσον αφορά τα δικαιώματα, η καθημερινή αποζημίωση και εκπατρισμό. Χρειάζεται και τεκμηριωμένη λογική που θα ακολουθείτε και θα πρέπει να καλυφθούν και ανεπάρκει όσον αφορά τα διάφορα απαιτούμενα έγγραφα που να χορηγούνται και συγκεκριμένε διαδικασίε που αφορούν ε, τα, ταξιδιωτική αποζημίωση κατά αποκομήν ε, και εκεί ίσως να υπάρχει πρόβλημα και να υπάρχει δυνατότητα για σφάλματα. Γι' αυτό ε, συμφωνήσαμε να υπάρξει ένα σημείο δράσεως με 20 σημεία που καλύπτει 12 τομείς σημαντικού κινδύνου και 8 μετρίου κινδύνου στόχος ε, του ελέγχου, ε, τομέα εξωτερικής μετάφρασης για την προμήθεια και εφαρμογή του μέτρων ήταν να δούμε η διαδικασία ανάθεση συμμορφώνεται με τους κανόνες και για την ορθή ε, χρηστή οικονομική διαχείριση και δεύτερον να διαπιστώσουμε κατά πόσο η εφαρμογή του πλαισίου και των διαφόρων συμβάσεων μετά στο πλαίσιο ελέγχονται αρκετά και να εξασφαλιστεί η τεχνική ποιότητα των μεταφράσεων και έτσι θα πρέπει να καλύπτονται με αυτόν τον τρόπο ενάγκε του Κοινοβούλιο. Έλεγχο επιβεβαίωσε ότι εστιάζεται σωστά η Γενική Διεύθυνση Μετάφραση και έτσι συμμορφούται η διαδικασία που ακολουθεί με του κανόνε και τι διατάξει περί αναθέσεων συμβάσεων. Επίση, βρήκε πεδίο να καλυφθούν κάποια προβλήματα μέσω πρώτα απ' όλα μέτρων, τόσο ώστε να βελτιωθεί η διοργάνωση τη διαδικασία διαγωνισμών συμπεριλαμβανομένη πιο έγκαιρου αιτήματο για συμπληρωματικέ πληροφορίε και να βελτιωθεί επίση η αξιολόγηση. Μετά χρειάζεται τα κριτήρια ανάθεσης να βελτιωθούν για την ποιότητα όσον αφορά τις μελλοντικού διαγωνισμούς. Τρίτον, μέτρα για να θεωρηθούν οι εξωτερικές εταιρείες να βελτιώσουν την ποιότητα των μεταφράσεων συμπεριλαμβανομένων ε, και μέσω ελέγχου εκ των υστέρων. Τέταρτον, θέλουμε να βελτιώσουμε την αξιοπιστία των υπολογισμών του πραγματικού πλήρους κόστους της εξωτερικής μετάφρασης. Για να καλυφθούν αυτά τα μέτρα, ο εσωτερικό έλεγχο συμφώνησε με ένα σχέδιο δράση με έξι σημεία με τη Γενική έθεση Μετάφραση. Δύο από αυτά τα σημεία αφορούν σημαντικό κίνδυνο και τέσσερα μέτριο κίνδυνο. Όσον αφορά το σύστημα πληροφοριών και τη σχετική στρατηγική του εσωτερικού ελέγχου, βασικό σκοπό ήταν να ελεγχθούν. Λοιπόν, σύμφωνα με τη στρατηγική για τα συστήματα πληροφορική. Βασικό στόχο ήταν ο έλεγχο των αποκεντρωμένων των δραστηριοτήτων της αποκεντρωμένης τεχνολογίας. Βασικός στόχος ήταν να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των αποκεντρωμένων συστημάτων πληροφορικής για το σχεδιασμό, την εκτέλεση, συντήρηση και υποστήριξη λύσεων πληροφορικής, εστιαζόμενοι επί δείγματος γενικών διευθύνσεων σε διαφορετικά επίπεδα οριμότητας και κλίμακας και δεύτερον εξολογηθεί ο ρόλος της Γενικής Διευθύνσεως ITEC όσον αφορά τις ε, επιδόσεις αποκεντρωμένων ε, λειτουργιών. Τι βρήκε ο έλεγχος, ότι εν γέννη η αποκέντρωση των αστυνομικών πληροφορικής προ τι γράφω γενικέ διευθύνσει βοήθησε να βελτιωθεί η ανταπόκριση στι απαιτήσει επιχειρησιακέ. Επίση, άλλο έβριμα ήταν ότι οι αποκεντρωμένε μονάδε σταδιακά ε, οριμάζουν αφορά τι επιχειρήσει του, χρησιμοποιώντα τα σχετικά πρότυπα και βέλτιστε πρακτικέ για τη βελτίωση, την εξέβρεση λύσεων και την παροχή αποτελεσματική υποστήριξη και συντήρηση. Για να πετευθούν τα πλήρη ωφέλη της αποκεντρώσεω, ο έλεγχος ενετόπισε πεδίο για κάλυψη των κάτω θεμάτων. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται ενίσχυση της, του ελέγχου του προϋπολογισμού που διατίθεται για πρωτοβουλίες για την πληροφορική, όσα αυτά συντονίζονται στα πλαίσια του προγράμματος IT για την πληροφορική. Δεύτερον, να αυξηθεί η βεβαιότητα ότι οι πρωτοβουλίες για την πληροφορική υλοποιούνται εγκαίρως για το συγκεκριμένο συμπεφωνημένο στόχο στα πλαίσια τη απαιτούμενη ποιότητα και εντό των χρημάτων που είχαν προβληθεί του θα πρέπει οι αποκεντρωμένες μονάδες να βελτιώσουν τον έλεγχό τους και την αξιολόγηση των νέων ε, εκδόσεων του λογισμικού και των ε, ε, διαφόρων προβλημάτων που διαχειρίζονται. Λοιπόν, θα πρέπει, θα πρέπει πρώτα απ' όλα σταδιακά να μετακινηθούμε και οι αναθέσεις των συμβάσεων να μετακινηθούν από μέσα και χρόνο που είχαν σαν πρώτη στο στόχο να πάμε στην τεχνογνωσία και τα αποτελέσματα. Συζητήσαμε με τι γενικέ διευθύνσει αυτά τα προβλήματα και ολοκληρώνονται οι συζητήσει για να καλυφθούν τα προαναφερθέντα προβλήματα. Το 2017 ο εσωτερικό έλεγχο ε, εξετέλεσε δύο αποστολέ διαβούλευση. Στα πλαίσια των επαγγελματικών προτύπων, αυτέ οι αποστολέ είχαν συμβουλευτική φύση κατόπιν αιτήσεων των διαφόρων γενικών διευθύνσεων και με συγκεκριμένο στόχο. Πρώτο στόχο ήταν η Γενική Διεύθυνση για την Επικοινωνία. Ε, ήθελε καινούργια νομοτολογία για τι όσον αφορά τον προπολογισμό ε, και αφορούσαν πολλά κονδύλια του προπολογισμού και μόνο κάποια κονδύλια είχαν συγκεκριμένη ε, σύνδεση με την επικοινωνία. Θέλαμε επικαιροποίηση ούτω ώστε η ονοματολογία να αντικατοπτεί την πραγματικότητα. Τα αποτελέσματα τη προσπάθεια ήταν ο εσωτερικό έλεγχο συμφώνησε και υποστηρίζει τι ε, αναθεωρήσει που πρότεινε η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνία. Για να βοηθήσουμε τη Γενική Διεύθυνση να τα εφαρμόσει όλα αυτά, ο εσωτερικό έλεγχο έκανε τι συστάσει όσον αφορά την παρουσίαση τη σύνταξη ενό επικοινωνιακού σχεδίου κάθε χρόνο, να εντοπιστούν οι διάφορες τεχνική φύσεω δαπάνε και να υπάρξει πλήρης αναφορά του, των ε, δαπανών. Η δεύτερη αποστολή που ήταν της ε, υπηρεσία ε, έρευνας του Κοινοβουλίου της EPRS αφορούσε την αγορά για τις, για τις εγγραφές σε συνδρομές σε, σε βιβλιοθήκες για να βοηθήσουμε την βιβλιοθήκη να βελτιώσει αυτή τη δραστηριότητα, κάναμε έξι συστάσεις. Πρώτα απ' όλα, να υπάρχουν προδιαγραφές για απόκτηση και ακύρωση στις, σύμφωνα με τους κανόνες των βιβλιοθηκών, να ξέρουμε οι τελικοί χρήστες ποια τι άποψη έχουν, να έχουμε στατιστικά στοιχεία για τη χρήση, να ταξινομηθούν οι χρήστες και τα προϊόντα και να παρέχονται κατά ζήτηση διάφορες υπηρεσίες ε, στα, αντί από κάποιες μακροπρόθεσμες εγγραφές. Λοιπόν, ε, θεωρούμε λοιπόν ποιες είναι οι ανοιχτές δράσεις, τις αξιολογούμε από τις προηγούμενες από τους ούγμους ελέγχους τι έχει γίνει μέχρι τώρα και κάθε χρόνο κάνουμε δύο τους ελέγχους, τι συνέχεια έχει δοθεί. Κάναμε δύο ελέγχους το 2017, αξιολογήσαμε 71 ανοιχτέ δράσεις και εσωτερικό έλεγχος μπόρεσε να κλείσει 34 από αυτές. Η πρόοδος πέντε άλλων δράσεων ε, μας οδήγησε να μειωθεί ο υποβόσκων κίνδυνος από σημαντική κίνδυνη γίνανε μέτρη και στην έκτη περίπτωση ο κίνδυνος αυξήθηκε από μέτριο σε σημαντικό. Έχουμε ανοιχτέ δράσει που αντιμετώπισαν σημαντικό ε, κίνδυνο και οι δράσει αυτέ από 26 έγιναν 11. Οπότε μειώνουμε γενικά τον, ε, τον κίνδυνο των ανοιχτών δράσεων, των εκκρεμώσεων δράσεων. Δεν υπήρχαν εκκρεμούσε δράσει στην κατηγορία του υψηλού κινδύνου. Ο έλεγχο του 2017 επίση συμπεριέλαβε το πρώτο τμήμα ενό ελέγχου στον τομέα τη συντηρήσεω των κτηρίων, ε, νέου εξοπλισμού και ανανέωση του εξοπλισμού, κάτι που συνεχίστηκε το 2018. Η εκθέση υιοθετήθηκε στις 12 Οκτωβρίου του 2018 και θα συμπεριληφθεί σαν ένα τμήμα των δραστηριοτήτων του 2018. Η ετήσια έκθεση περιγράφει την εφαρμογή της δικής του ποιοτική, ποιοτικού ελέγχου και της βελτιώσεως του προγράμματος. Σύμφωνα με τα πρότυπά μα, κάθε υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να υποστήξει εξωτερική αξιολόγηση από ειδικό ε, εξωτερικό φορέα κάθε πέντε χρόνια. Η εξορίση του 2016 οδήγησε ε, στον εξωτερικό αξιολογητή να δείξει ότι ο εσωτερικό έλεγχο λειτουργούσε στα ύψιστα πρότυπα. Σύμφωνα με τι διαγραφές. το πρόγραμμα του 2017 εστιάστηκε για περαιτέρω βελτίωση. Στο τμήμα 4 τη εκθέσεω περιγράφεται ο ρόλο ε, του πάνελ του ελέγχου που ελέγχει τον κίνδυνο και ελέγχει οι αιτικές διαδικασίες που χειρίζεται η διοίκηση και εξηγεί πώς η δομή του πάνελ και η λειτουργία του πάνελ συνάδουν με τη βέστητη πρακτική στη διακυβέρνηση επιχειρήσεων. Στο, στο τρίτο τμήμα έχουμε τα συμπεράσματα της εκθέσεως και εξηγούμε πώς η δραστηριότητα του 2017 εστιάστηκε στην παροχή της διαβεβαίωσης συμμορφώσεως με την αρχή της ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης και πιο συγκεκριμένα την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της διαχείρισης, διαχείριση του κινδύνου και τις ελεγκτικές διαδικασίες σε διάφορους τομείς. Ε, τέλος, εσωτερικός ελεγκτής επιβεβαιώνει ότι η ανεξαρτησία του δεν επιβεβαιάστηκε ότι υπονομεύτηκε το 2017. Εν κατακλείδη, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του ελεγκτικού πάνελ και το Γενικό Γραμματέα για την υποστήριξή του και τι συμβουλέ που έδωσαν το 2017 και να εκφράσω την εκτίμησή μου για την έξοχη συνεργασία που ε, επεδείχθη έναντι των διαφόρων τμήματων της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Η συγγήτρια κυρία Σμίτ έχει το λόγο για την πρώτη ε, ανταλλαγή απόψε. Ευχαριστώ. Μετά από τόσο έπαινο για το Γενικό Γραμματέα, εγώ θα ήθελα να παίξω τον αντίθετο ρόλο, αλλά ε, που είναι δύσκολο. Πρέπει να σας πω ότι έχω συναντήσει διάφορες γενικές διευθύνσεις γιατί θέλω να έχω ίδια εικόνα και να τα βλέπω με τα μάτια μου. Όλοι δήλωσαν προθυμία να με συναντήσουν και να απαντήσουν και στις ε, επικριτικές ερωτήσεις, καμιά φορά και σε ανόητες ερωτήσεις που τους έκανα. Πραγματικά όπου και να πήγα που πήγα σχεδόν σε όλες τις γενικές διευθύνσεις. Ήταν ανοιχτή και ειλικρινή στη συζήτηση. Πολλά πράγματα τα οποία ε, ρώτησα ε, ή αμφέβαλα από την προηγουμένη μου εμπειρία ε, τα έθεσα και τουλάχιστον με άκουγαν πάντα και μου απαντούσαν. Ας πούμε, ήθελα να δω όλα τα γραφεία και να πω και στο τελευταίο υπόγειο και στο ε, τελευταίο πατάρι ε, και παντού ε, διαπίστωσα ότι κανείς ε, δεν είχε να κρύψει τίποτα, δεν ήθελε να κρύψει τίποτα και γίνεται προσπάθεια πάντα για ειλικρινή και ανοιχτή συνεργασία. Και εγώ έχω μεγάλο έπαινο και παρακαλώ να τα διαβιβάσετε. Εκεί λοιπόν που τα ανακάτωνα όλα και τα έψαχνα, και τα ψήριζα, ε, έπεσα και σε κάποια πράγματα που δεν ήταν πάντα ε, καλά και άγια ε, και που μας δημιουργούν προβλήματα και σκέψεις. Όλη αυτή η ιστορία με την ασφάλεια. Καλό είναι που τώρα εξασφαλίζονται τα κτίρια και προστατεύονται καλύτερα και είναι καλύτερος ο εξοπλισμός, αλλά εγώ ως μεμονωμένη βουλευτής και μετά από όσα άκουσα και από άλλους συναδέλφους, από βοηθούς και νομίζω ότι δεν υπάρχει μια πολύ αυστηρή στρατηγική ασφαλείας που να την ε, βλέπουμε κιόλας. Παρόλο που είμαστε σε επίπεδο ασφαλείας κίτρινο, μπορεί κάποιος να μπει στον καράζ χωρίς να έχει το σήμα το, το, την κάρτα ο ίδιος ή το αυτοκίνητο. Και να μην το σταματούν, ακόμα και αν μεταφέρει κάποια πράγματα. Αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να ελέγχεται αυστηρά και ανησυχώ λίγο για ε, αυτή τη μάζα των επισκεπτών που κυκλοφορούν στο κοινοβούλιο. Ξέρω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι διαπιστευμένοι και τα λοιπά, αλλά έχουμε γεμίσει επισκέπτε εδώ πέρα, όχι μόνο στο Στρασβουργό και στι Βρυξέλλε. Μου φαίνονται λίγο περίεργα αυτά. Και μετά όλη αυτή η ιστορία που με ενδιαφέρε πάρα πολύ ήταν η υπηρεσία των οδηγών και οι διαφορές, ε, η μετάβαση τώρα σε υβριδικά οχήματα και ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα ή η πρόσληψη ε, οδηγών που είναι υπάλληλοι του Κοινοβουλίου. Νομίζω το έχω πει ε, επανειλημμένα και ρώτησα και πολλές φορές. Έχει βελτιωθεί ε, η κατάσταση από τότε που έχουμε δικούς μας υπαλλήλους και τώρα ε, πραγματικά μπορούμε να ελέγχουμε καλύτερα την κατάσταση. Και οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ φιλικοί, ευγενικοί, δεν έχω κανένα πρόβλημα και κανένα αρνητικό ε, να πω. Ένα άλλο ερώτημα μου γεννήθηκε όταν μπήκα για πρώτη φορά στο κοινοβούλιο πριν από πέντε χρόνια είναι όλα αυτά που έχουμε, που είχαμε σούπερ μάρκετ, γυμναστήριο, καθαριστήριο κτλ. Ε, ε, τώρα το σούπερ μάρκετ έκλεισε. Τι θα γίνει, θα ξανανοίξει, θα πάει κάπου αλλού, γιατί δεν είναι καθόλου ε, ασήμαντα αυτά τα πράγματα που έχουν να κάνουν και με την ασφάλεια στα κτίρια μας. Και μας χρειάζονται αυτά, είναι άχρηστα. Τεράστια προβλήματα είχα επίσης ε, με ε, τα θέματα της ε, πληροφορικής. Όπως και πολλοί συνάδελφοι, εγώ χρησιμοποιώ συσκευές Apple και πολύ συχνά βρίσκω τα όρια μου. Ε, δεν μπορώ να διαβάσω τα mail μου στο iPad ή στο iPhone. Ε, γιατί χρειάζεται καμιά φορά εκτυπωτής και πού να το βρω τον εκτυπωτή και τα λοιπά. Ε, έχω πρόβλημα με την πληροφορική και την επικοινωνία, το ICT. Ξέρω ότι για να είσαι πληροφορικάριος πρέπει να το έχει. Ε, εντάξει, αλλά θα πρέπει να έχουν και μια στοιχειώδη υπηρεσία την οποία να παρέχουν στους πελάτες. Και ε, καλό θα ήταν να εκπαιδεύονται και εκεί οι υπάλληλοι. Γιατί το πρώτο που σου λένε, α, όχι, αυτό δεν γίνεται, αυτό δεν επιτρέπεται, αυτό δεν κάνει. Ε, ε, τώρα έχουν βελτιωθεί τα πράγματα ε, πέρα από τους υβριδικούς υπολογιστές και ε, την ιστοσελίδα. Υπάρχει χώρος ε, για βελτίωση και πεδίο δράσης και ενώπιση των εκλογών όπου πολλά πράγματα είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι τα γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Αυτά. Αυτά τα σκέφτηκα ε, την ώρα που μιλούσατε και δεν τηρώ αυτά που έχω γράψει εδώ. Ε, το ποσοστό σφάλματος είναι καταπληκτικό και απαντήσατε και σε 161 ερωτήσεις που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη προσπάθεια και μάλιστα η απάντηση ήταν πάρα πολύ εμπεριστατωμένη και αυτή και καταβάλλατε κόπο. Πολύ ωραία πράγματα. Κάποιες λεπτομέρειες όμως υπάρχουν ε, που ανέκυψαν απαντώντας σε κάποια ερώτηση για τα γραφεία συνδέσμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις διάφορε πρωτεύουσες και στα κράτη-μέλη. Ας πούμε, όταν εγώ είμαι εισηγήτρια, ε, μπορούν να προσκαλούνται εκεί ενδιαφερόμενοι και να με στηρίζουν στην πολιτική νομοθετική μου δραστηριότητα. Δεν ξέρω, σε άλλες χώρες αυτό μπορεί να ισχύει στη δική μου χώρα καμία σχέση. Δεν το έχω ζήσει ποτέ στη ζωή μου, δεν είχα αυτή την ευτυχία. Δεν ξέρω, γίνεται κάποιος έλεγχος εκεί υπάρχει κάποια σαφής περιγραφή της κατάστασης. Εγώ φταίω μήπως παρέλειψα να ρωτήσω, να το ζητήσω. Πώς έχει η επικοινωνία με τους βουλευτές. Πρέπει εκείνοι να τη ζητήσουν, πρέπει να τους παρέχεται η υπηρεσία. Και τι γίνεται με τα δύο γραφεία που έχουμε τώρα συνδέσμους στο Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνουν για τη μεταβατική περίοδο ή θα κλείσουν αμέσως, πώς θα γίνει αυτό. Και άλλη μια ερώτηση. Ακούσαμε ότι κάποια από τα αντικείμενά μας τα αγοράζουμε, ε, κάποια τα νοικιάζουμε, ε, έχουν και τα υπέρ και τα κατά. Πώς γίνεται αυτό, γιατί υπάρχει το θέμα της συντήρησης, δεν μιλώ μόνο, για τα κτίρια, ε, ε η πρόεδρος ε, μου ε, υποδεικνύει το χρόνο, αλλά θέλω λίγο χρόνο. Υπάρχει μια στρατηγική. Και απαντώντας στις ερωτήσεις, επίσης, αναφερθήκατε στο αγαπημένο θέμα του συνταξιδοτικού ταμείου. Είχα και εγώ λιλογραφία με τον πρόεδρο, του Ταμείου. Υπάρχει καμιά ιδέα εκεί καινούργια. Έχω πολλές άλλες ερωτήσει. τώρα δεν τολμώ, γιατί η πρόεδρος μου δείχνει το ρολόι. Τι να κάνω, ευχαριστώ. Υποδειγματικοί είσαστε. Κύριος Γενικός, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς, ασφάλεια έγινε λόγος για την ελεύθερη κυκλοφορία των ομάδων επισκεπτών στο κτίριο. Προσπαθούμε με την ε, καθίδρυση νέων ε, εγκαταστάσεων, ε, εννέα των αριθμών, να έχουμε έχουν, των νέων μάλλον εγκαταστάσεων να είναι απομονωμένες αυτές από το υπόλοιπο κτίριο όπως το Παρλαμεντάριουμ, όπως το ο οίκος Ευρωπαϊκής Ιστορίας, όπως οι νέες εγκαταστάσεις του Άτριουμ που ακόμα βέβαια χρησιμοποιούνται για τα ε, τουριστικά λεωφορεία ε, θα συνδεθεί στη συνέχεια με τις ε, αίθουσε όπου θα γίνονται οι παρουσιάσει, αλλά θα είναι απομονωμένο όπως και τα προηγούμενα από τα λειτουργικά μας κτίρια το... ο σταθμός, το ίδιο, το InfoPoint που θα ανακαινιστεί την επόμενη διετία, απομονωμένο από, το κεντρικό, από τα κεντρικά κτίρια, από το συνολικό κτίριακό μας ε, ε, συγκρότημα. Δηλαδή βήμα-βήμα περνούμε στην κατάσταση όπου θα έχουμε ένα χωριστό δρομολόγιο σε για τους ε, επισκέπτες που έτσι δεν θα περνούν μέσα στο κυρίως κτίριο. Θα υπάρχει ειδική είσοδος για τους ε, ε, επισκέπτες που όμως δεν θα έχουν πρόσβαση στο γενικό κτίριο, στο, στο κτηριακό μας συγκρότημα. Και μετά θα είναι πολιτική η απόφαση το να αποφασίσουν οι βουλευτές ότι έχουμε παραδείγματι την εκδήλωση τάδε, ε, δίνα, 60.000 στο Station Europe, 150 στο κέντρο, στο Νίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, όλους αυτούς τους επισκέπτες λοιπόν, ε, αποφασίζεται ή θα αποφασιστεί πολιτικά να ε, μην έχουν πρόσβαση στα κτίρια. Μια αλλαγή νοοτροπίας ίσως, μια, μια πολιτική απόφαση πάντως που θα πρέπει να ληφθεί για να υλοποιηθεί αυτό. Πάντω τη δυνατότητα θα την έχουμε να μην έχουν πρόσβαση οι επισκέπτε. Είμαστε πολύ κοντά δηλαδή σε, ε, στη, ε, στάδιο κοινό της προετοιμασίας που θα είμαστε σε θέση να πούμε ότι να, και δεδομένη τη κατάσταση σχετική με την ασφάλεια οι ε, επισκέπτες δεν θα μπαίνουν στα κτίρια, ε, του, στα κτίρια του Κοινοβούλου, αλλά θα πρέπει να ληφθεί μια πολιτική απόφαση, όπως είπα του Προεδρείου. Ασφάλεια τώρα τον κύριο εξωτερική ασφάλεια. Τα τελευταία δέκα χρόνια έχουμε διανύσει πολύ δρόμο. Η κατάσταση ήταν στο παρελθόν ότι γενικά όταν είχαμε θέμα ασφάλειας δεν φαινόταν πολύ ευπρόσδεκτο ε, και γενικά είχαμε την ε, τάση να έχουμε κλίμα ανοιχτό, πνεύμα ανοιχτό στους ξένους κτλ. Αλλά ήρθαν οι μέρες όπου 200 Κούρδοι κάναν εισβολή στο κτίριο, έγιναν μετά και οι ε, τρομοκρατικές επιθέσεις, εκ των οποίων η μία αφορούσε τον σταθμό του μετρό που χρησιμοποιούμε το δικό μας το προσωπικό. Και ήταν θαύμα το ότι έλαβε χώρα τόσο νωρί που δεν είχαμε δικούς μας υπαλλήλου μεταξύ των θυμάτων, εκτός από έναν σταζιέχ, παρανασκούμενο. Όλα αυτά λοιπόν τα γεγονότα μας υποχρέωσαν να αντλήσουμε τα διδάγματα, να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες ε, και να κάνουμε τις σχετικές διορθώσεις. Παραμένουν κρεμή βέβαια ζητήματα όπως ε, η εισαγωγή ενός ε, badge, μιας κάρτας εισόδου που δεν θα μπορεί να πλαστογραφηθεί, αλλά και θέμα το οποίο έχει μάλιστα αρκετά έντονα στο Προεδρείο για το αν ορισμένα οι του κτηρίου θα είναι απομονωμένοι, δεν θα έχουν πρόσβαση δηλαδή οι πάντες, γιατί είδαμε κάποιες ε, περιπτώσεις όπου κάποιοι άσχετοι μπήκανε μέσα στο γραφείο ενός ε, βουλευτή απρόσκλητη. Είναι ζητήματα τα οποία έχουν συζητηθεί τα τελευταία χρόνια υπό τον τίτλο ε, zoning, δηλαδή περιορισμό ε, πρόσβαση σε ορισμένε ζώνε του κτίριου. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφασίσει το Προεδρείο. Ευχαριστώ πολύ για την θετική αξιολόγηση για την υπηρεσία των οδηγών. Βεβαίως και η γεωγραφική κατανομή έχει μεγάλη σημασία. Βλέπουμε ποια είναι τα κράτη που έχουν μεγαλύτερη εκπροσώπευση στην υπηρεσία αυτή. Πάντως, είναι γενικά θετική οι αντίκτυποι που λαμβάνουμε και από τους βουλευτές, μάλιστα έγινε και μια αξιολόγηση που παρουσιάστηκε στο Προεδρείο και εν γέννη το Προεδρείο αποφάσισε ότι παρότι ήταν κάπως διαφιλονικούμενη η εισαγωγή του μέτρου του, της υπηρεσίας και σε επίπεδο ολομέλειας, ότι ήταν τελικά ε, πολύ καλή επιλογή. Έχει γίνει επαλήθευση και σε όρους ασφαλείας των διαπιστευτηρίων των ε, υπαλλήλων αυτών υπάρχει γενικά τέτοιο σύστημα ασφαλείας και στην πρόσβαση στα γκαράζ μας που δεν ε, μπορεί να γεννηθεί πρόβλημα ασφάλειας. Επίσης, Για το θέμα του σούπερ μάρκετ είπατε ότι και εσείς μπορεί να αλλάξατε κάπως στάση σε σχέση με την πρώτη σας εντύπωση όταν ήρθατε. Βεβαίως βολεύει να μπορούμε να κάνουμε κάποια ε, μικροαγορά, κάποια ψώνια που χρειαζόμαστε γρήγορα και το ε, γυμναστήριο βεβαίως. Αν και θεωρώ προσωπικώς ότι έχει μεγάλη σημασία να είναι διαθέσιμο και τόσο για τους βουλευτές όσο και για το προσωπικό. Πληροφορική. ICT. Πάντα πρέπει να εξισορροπούμε την ανάγκη της ε, δυνατότητας εξυπηρέτησης του χρήστη με πνεύμα ανοιχτό, αλλά και της προστασίας της ασφάλειας του συστήματος. Μια στάθμιση λοιπόν πρέπει να γίνεται πάντα, γιατί μέχρι τώρα δίναμε μεγάλο βάρος στην ασφάλεια και ως εκ τούτου δεν είδαμε σοβαρά επεισόδια ως προς την ασφάλεια της χρήσης της πληροφορικής, αλλά στο μπορούσαμε και στην εξυπηρέτηση των χρηστών να βελτιωθούμε γιατί ε, γιατί τις είδαμε και από την προηγούμενη θητεία πως υπήρξαν οι εισηγητές που επεδίωξαν ε, διάλογο όχι στην ε, οικία χώρα αλλά σε άλλη χώρα διάλογο με τους ε, εμπλεκόμενους φορείς όπως λέμε και άρα ο διάλογος δεν έλαβε χώρα απαραίτητα στις Βεξίλες στο Στρασβούργο αλλά και σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τέτοιου είδους εκδηλώσεις καλύπτονται τα, τα έξοδα από τον προϋπολογισμό πλέον δεν πρέπει να τα αναλάβει ο βουλευτής μόνος του. Και βεβαίως να πρόκειται για έκθεση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ε, το Προεδρείο θα την υποστηρίξει. Για τα γραφεία μας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οριστική απόφαση δεν υπάρχει. Ωστόσο, το Προεδρείο έχει ξεκινήσει τη συζήτηση. Το γραφείο του Λονδίνου, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ από αυτές τις συζητήσεις, διατηρείται ώστε να διαφυλαχθεί και αυτή η στενή σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και για να μην χάσουμε την δυνατότητα υποστηρίξη των τριών εκατομμυρίων ε, ε, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι κατεστημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για το Εδιμβούργο θα πρέπει το Προεδρείο να λάβει απόφαση για το γραφείο του Εδιμβούργου, η οποία πάντως ε, απόφαση δεν θα τεθεί σε εφαρμογή ε, πριν από το πέρας της μεταβατικής περίοδου, δηλαδή πριν τα τέλη του 2020 όπως έχουν τώρα τα πράγματα και άρα και το σχετικό προσωπικό παραμένει εκεί, ε, δεν επηρεάζονται ούτε συμβάσει τους, ούτε τίποτα, ούτε οικογενειακή του ζωή. Για την αγορά ή την, εκμίστοση, την μίσθωση κτίριων. Η προτίμησή μας είναι προς την αγορά πάντα, με βάση και έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου χρόνια πριν, που έλεγε ότι θα πρέπει η επιλογή να τίνει προς την αγορά ακινήτων αυτό και ε, πράξαμε. 90% έχουμε, ε, τα κτίρια που χρησιμοποιούμε είναι ιδιόκτητα. Βεβαίω υπάρχει σχετική επιβάρυνση για την ανακαίνιση τους ε, που μας επιβαρύνει, που μας αντιστοιχεί. Ε, βεβαίως θα πρέπει να δούμε και πού υπάρχει δυνατότητα να αγοραστεί ένα κτίριο εάν πρόκειται παραδείγματι για γραφείο ενημέρωση κοινού και αν τυχόν στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν προσφέρεται προς αγορά, τότε μισθώνουμε. Για το Στεξιωτικό Ταμείο που ανέφερε ήδη και τοποθετήθηκε ο Αντιπρόεδρος κ. Σασόλη, το Μάρτιο στο Προεδρείο είχα κάνει τη σχετική πρόταση και το Προεδρείο εξέφρασε την επιθυμία για άλλη μια φορά να ασχοληθεί με το θέμα αυτό το νομική υπηρεσία, αλλά και ταυτόχρονα να ε, μελετηθεί πολύ πιο προσεκτικά το ιστορικό αυτού του εξωτικού Ταμείου. Ε, τα δύο αυτά, οι δύο αυτές προϋποθέσεις έχουν το μεταξύ πληρωθεί και έτσι σύντομα, δηλαδή κάπου τον Δεκέμβριο, πρόκειται να ασχοληθεί το Προεδρείο γιατί έχει αποφασίσει ο Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος είναι εκείνος ο οποίος ορίζει την ε, ημερήσια διάταξη του Προεδρείου. Διάφορες επιλογές έχουμε στη διάθεσή μας ε, η κάθε μια από αυτές παρουσιάζει συγκεκριμένους κινδύνους ως προς τα νομικά ζητήματα και με βάση τη στάθμιση στην οποία θα προβεί το, το Προεδρείο θα λάβει και την απόφαση της επιλογής του σχετικού μέτρου για τον περιορισμό του ελλείμματος του εξωτικού ταμείου. Ευχαριστώ. Και τώρα ακολουθούμε σκιώδης, παρακαλώ, σύντομα. Μετά από τέσσερα λεπτά θα σας διακόπτω. Η κυρία Γιάλα Σέντερ πρώτη, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος του συναδέλφου Παχνιό θα μιλήσω. Είναι αρμόδιος και όδης ηγετής, αλλά δυστυχώς κολλείεται για λόγους ανελημμένων υποχρεώσεων να συμμετέχει στη σημερινή συνεδρία. Βλέπω ότι στην περίπτωση της απαλλαγής χρησιμοποιήθηκε αυτό το help desk και θέλω να ρωτήσω και τον κύριο Γκάλβεν και την κυρία Κλάουντια Σμιτ, γιατί βλέπω ότι έχει δημιουργηθεί έτσι μια υπηρεσία για να μας ε, βοηθάει. Δεν ξέρω, σας βοηθάει και σας κύριε Γκάλβιν, εντάξει αστείευομαι. Κανονικά για την απαλλαγή δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα ε, με τις γενικές διευθύνσεις επικοινωνούσαμε και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Τώρα γιατί φτιάξατε υπηρεσία που χρειάζεται να βοηθάει τους βουλευτές, ε, τους συγγητές, ε, πόσους υπαλλήλους απαρτίζεται και υπάρχει κανένα πρόβλημα σύγκρουση συμφερόντων. Αν το έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήμασταν έξαλλοι τώρα. Επίσης, ε, για το Προεδρείο, πώς εργάζεται, πώς λαμβάνονται αποφάσεις, πώς εφαρμόζονται, πώς ε, παρακολουθούνται και πώς αξιολογούνται στην εφαρμογή τους, γιατί εξακολουθούμε να έχουμε προβλήματα με τη διαφάνεια προς τη διαδικασία. Καμιά φορά όταν ε, ζητούμε ε, ε, από το Γενικό Γραμματέα να μας απαντήσει, μας παραπέμπει στο Προεδρείο. Μα για να απαντήσει το Προεδρείο χρειάζεται μια προεργασία και μετά ο Γενικός Γραμματέας εφαρμόζει και παρακολουθεί την υλοποίηση αυτής της εφαρμογής. Και θέλω να μου το διευκρινίσετε. Ε, απολαβές και συντάξεις των, συντα... των διαπιστευμένων βοηθών. Τι γίνεται με τα συνταξιοδιατικά δικαιώματα εκείνων που δεν συμπληρώνουν 10 χρόνια. Οι πολιτικές ομάδες δείχνουν μια αλληλεγγύη. Η εργατική αλληλεγγύη κιόλας. Έχουν δικό τους καθεστώς οι διαπιστευμένοι βοηθοί. Και η λύση θα πρέπει να είναι θεσμική. Και να μην ζητάνε μη ζητάτε από τα, τις πολιτικές ομάδες να λύσει ένα πρόβλημα που το, το πρόβλημα αφορά όλο το κοινοβούλιο. Εντάξει, μπορεί ο κάθε βοηθός να είναι βοηθός ενός βουλευτή, αλλά υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο. Και για τις συντάξεις λέτε ότι δεν έχουν υπογράψει εγκαίρον τις συμβάσεις ή δεν τις έχουν συμπληρώσει εγκαίρως. Ενώ εμεί γνωρίζουμε ότι δεν ήταν σε θέση η διοίκηση να διαχειριστεί όλη αυτή τη πληθώρα και τον όγκο των συμβάσεων. Συγγνώμη. Η επίρρηψη ευθυνών, οι αλληλοκατηγορίε δεν λύνουν το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι θεσμικό, άρα θα πρέπει θεσμικά να λυθεί από το Κοινοβούλιο. Και ο κάθε κανονίζει την πορεία του, αλλά να μην τα ρίχνει ο ένα τον άλλον. Γιατί τελειώνει η θητεία και λύση δεν θα έχουμε. Το ίδιο για τις απολαβές των βοηθών ε, και την ε, ημερήσια αποζημίωση. Ε, υπάρχει μια πολύ ειδική ρύθμιση χωρίς αναδρομική ισχύ όπως για το υπόλοιπο προσωπικό και τους υπόλοιπους υπαλλήλους. Είναι λίγο προβληματικό αυτό. Και σε σχέση με τα γραφεία βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον το 2019 και παρακαλώ να μου το διευκρινίσετε. Στο Στρασβούργο θα έχουμε ένα γραφείο για το βουλευτή και ένα γραφείο για τους βοηθούς. Πώς θα γίνει αυτό και πώς θα το εφαρμόσετε. Μετά, για τη χρήση των αυτοκινήτων, όλο και περισσότερο, τουλάχιστον σε μένα μου είχε αυτό τελευταία, να μοιραζόμαστε τα αυτοκίνητα με γενικού διευθυντέ. Τελείωσε ο χρόνο σα, τέσσερα λεπτά. Α, καλώ, μάλιστα, ναι. Εντάξει. Γραπτό θα συνεχιστεί η αλληλογραφία με το Γενικό Γραμματέα και θα μας απαντήσει. Κρίμα που δεν μπορούμε να το κάνουμε δημόσια εδώ. Ο κύριος Αλή, επόμενο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Σμιτ, αγαπητέ και σας όλοι, κυρία Βέλε, κύριε Γκάλμεν, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ καταρχάς για τις λεπτομερείς απαντήσεις που δόθηκαν στις ερωτήσεις μας. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του Ευρωκοινοβουλίου για το 2017. Η χρήση των οικονομικών πόρων για την επίτευξη στόχων του έτους. Τα αποτελέσματα άκουσαν ενθαρρυντικά. Το 2017, όπου είχαμε ένα δις 910 εκατομμύρια ευρώ, μόνο 0,9% έπρεπε να κυρωθούν από τα χρήματα αυτά του προπολογισμού. Αποδειχνεί την πολύ καλή διαχείριση των οικονομικών πόρων. Το είπε αυτό άλλωστε και ο Σασόλη. Οι στόχοι και τα αποτελέσματα του έτους απορρέουν από τις θεθείς προτεραιότητες από τους φορείς του Κοινοβουλίου που προετοίμασαν, κατάρτισαν τον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2017. Κάποια συγκεκριμένα θέματα να θέσω. Πρώτο, κάτι σημαντικότατο για τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμού. Η τεχνογνωσία για λογιστικά και έλεγχο που πρέπει να βελτιωθούν εντός του Κοινοβουλίου και στα πλαίσια της προετοιμασίας για την έκθεση απαλλαγής. Βελτιώθηκε το εσωτερικό σύστημα ελέγχου και της γραμματείας. Δεύτερον, δώσατε λεπτομερείς πληροφορίες τη λειτουργία του οίκου Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Είχαμε διάφορα προβλήματα στην Ένωση και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πόρους πολύτιμους για να προωθήσουμε καλύτερα την κατανόηση ευρωπαϊκής ιστορίας και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Από αυτή την άποψη, οι αριθμοί των επισκεπτών θα μπορούσαν να αυξηθούν μέσω εκστατείας ενημέρωσης. Τρίτον, για την αύξηση των προβλημάτων έχουμε τη μονάδα συμμόρφωσης που αναφέρεται στο Γενικό Διευθυντή της Υπηρεσίας Οικονομικών Θεμάτων. Στηρίζουμε την προσέγγιση για την αποφυγή ατασταλιών. Πώς μοιράζεται με την Επιτροπή μας αυτή η μονάδα της πληροφορία και τα, οι δυσκολίες οι τυχόν, πώς θα ξεπεραστούν. Τέλος. Συγχαρητήρια στην ηγεσία του Ευρωκοινοβουλίου για την καλή διαχείριση, διότι πέρσι υπήρξαν πολλά προβλήματα. Κυρίως όσον αφορά την ασφάλεια και όχι μόνο αυτό. Ξανά Συγχαρητήρια για αυτή την άριστη συμπεριφορά των αρμοδίων φορέων. για... Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε. Τρία σύντομα ερωτήματα. Το πρώτο, για τις γενικές δαπάνες και τα σχετικά κονδύλια, ο Αντιπρόεδρος σας όλοι το ανέφερε ακροθυγός. Θέλω λεπτομερέστερες εξηγήσεις Πότε θα ολοκληρωθούν οι σχετικές διαπραγματεύσεις. Από ό,τι ξέρω, δεν έχει επιτευχθεί η συμφωνία μεταξύ του Προεδρείου του Κοινοβουλίου και της αρμόδιας ομάδας για τον κανονισμό το σχετικό. Πότε θα ολοκληρωθούν οι εργασίες, πότε θα υπάρξει κάποια συμφωνία Προεδρείου και της ε, ομάδας μελέτης. Και όσον αφορά τι αποζημιώσει, σύμφωνα το άρθρο 62 των εφαρμοστικών μέτρων για το καταστατικό των μελών. Στο τέλος της θητείας, τα ποσά που δεν χρησιμοποιήθηκαν πρέπει να επιστραφούν από τις αποζημιώσεις. Υπάρχουν κάποια σχέδια από το Κοινοβούλιο να δοθούν τα κατάλληλα κριτήρια για την συμμόρφωση και για τις αποζημιώσεις αυτές. Σύμφωνα με τον κανονισμό, αυτά πρέπει να κρατούνται σε ένα ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό. Τι προβλέπετε για το σχετικό έλεγχο και να δώσουν πληροφορίε σε ευρωβουλευτέ για την κυβερνοασφάλεια μετά, για ενόψη των ευρωεκλογών. Υπάρχουν τεράστιε απειλέ. εναντίον των ευρωεκλογών. Μπορεί να απειληθούν ευρωεκλογέ από εξωτερικέ δυνάμει μέσω κυβερνοεπιθέσεων, μέσω ψευδών ειδήσεων και εκστρατιών παραπληροφόρηση. Μαζί με τα άλλα θεσμικά όργανα, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι σχέδια υπάρχουν, το Κοινοβούλιο τι θα κάνει για να αποφευθεί αυτό, τι θα γίνει για να υπάρξει προστασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από ψευδείς ειδήσει, κυβερνοεπιθέσεις, και παραπληροφόρηση. Μετά το νομοθετικό ίχνος. Συμφωνήθηκε να δημιουργηθεί δυνατότητα στην ιστοσελίδα του Ευρωκοινοβουλίου να μπορούν οι προβουλευτές να δημοσιεύουν εκθέσεις για το νομοθετικό ίχνος. Δεν είδα να υπάρχει ακόμα αυτή η δυνατότητα στην ιστοσελίδα. Αυτή η δυνατότητα που βρίσκεται αναμένεται σύντομα να υλοποιηθεί. Να μπορούν να δημοσιεύονται τα νομοθετικά ίχνη των εκθεσεών μας στην ιστοσελίδα. Συνάδελφε Ντεγιόγκ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, θα, θα ξεπεράσω το χρόνο μου. Ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις που μας δώσατε και τις προφορικές και τις απαντήσεις ε, στις ερωτήσεις μας. εν ώψη των ευρωεκλογών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ cool και πάρα πολύ in, αλλά τι γίνεται με την προεκλογική εκστρατεία και τις σχέσεις με τη νέα γενιά. Είναι μεγάλο ρίσκο, το θέσαμε και υπόψη του Προεδρείου και θα το προωθήσει, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ε, μπορούν ε, να ε, έχουν ε, πρόσβαση σε αυτή τη σούπερ προεκλογική εκστρατεία που κάνουμε. Είναι οι φτωχοί, οι άνθρωποι που θεωρούν ότι είναι όλο και πιο αποκλεισμένοι από το ευρωπαϊκό γίγνεσθε, γιατί δεν φτάνουμε σε αυτούς και θα ήθελα επίμονα να ρωτήσω και τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα τι θα γίνει διευρύνεται αυτή την εκστρατεία ενημέρωσης, να μην αφορά μόνο τους νέους και τους φοιτητές, γιατί θα πάνε όλα στραβά στις εκλογές. Στη συνέχεια υπάρχει κάποια αναντιστοιχία ε, των όσων ε, εμείς αποφασίζουμε για την ε, απαλλαγή και τις αποφάσεις του Προεδρείου. Μερικά πράγματα πηγαίνουν καλύτερα με τις καινούργιες ιστοσελίδες, που μπορούμε να συνδέσουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την προσωπική μας ιστοσελίδα, αλλά ε, ρωτώ πόσες πληροφορίες δίνονται στους ευρωβουλευτές. Και την ίδια ερώτηση έχω για το νομοθετικό ίχνος. Ε, γιατί ε, δεν μας έχει πει η Γενική Γραμματεία μερικά πράγματα για ε, τα ε, έντυπα όπου ανακοινώνουμε τη σχέση μας με τους λομπίστες. Ο Γενικός Γραμματέας κάνει πολλές προσπάθειες. Αλλά ε, Επίση, τι γίνεται, γιατί έχετε φαγωθεί να αντικαταστήσετε τον εξοπλισμό των γραφείων. Ε, δεν έχει ε, φθαρεί, είναι εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα αντικατάσταση. Τι γίνεται με τον οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Πόσα πληρώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για κάθε μέλος, για κάθε εργαζόμενο εκεί στο σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Υπάρχουν και κάποια προβλήματα με το προσωπικό. Ε, πώς αξιολογείτε τους υπαλλήλους. Ε, θα, έχουμε νέες ε, στολές για ε, ε, το προσωπικό ασφαλείας. Και όταν συζητάμε τις συντάξεις, χρησιμοποιείτε την Ισομερή Επιτροπή 200 και επίσης ε, ε, το προσωπικό του Μουσείου του Οίκου της Ευρωπαϊκής Ιστορίας ε, έχει το μισό μισθό από ότι ένα μεγάλο μουσείο στην Ολλανδία. Ο κύριος Γκερμπράντη. Ευχαριστώ. Κύριε Γενική Γραμματέα, κυρία Πρόεδρε, συγκεκριμένη ερώτηση έχω που συνδέεται με γραπτή ερώτηση την υπαριθμών 129 περί συνταξιωτικού ταμείου. Ρωτήσαμε για τη νομική βάση του συνταξιωτικού ταμείου. Ένας ειδικό για τα συνταξιωτικά μου είπε ότι το εθελοντικό αυτό συνταξιωτικό ταμείο τελικά είναι ιδιωτικό επενδυτικό μέσο μέτρα του Λουξεμβούργο και δεν υπάρχει λόγος η εσδήποτε νομική υποχρεώση από Κοινοβουλίου δεν υπήρχε τέτοια υποχρέωση να καταβάλει συντάξει. όταν η αναμενόμενη, η πραγματική αξία του ταμείου είναι χαμηλότερη το αναμενόμενο. Απάντηση λοιπόν, ποιο είναι το νομικό καθεστώς του ιδιωτικού αυτού επενδυτικού μέσου με έδρα το Λουξεμβούργο. Η πρόεδρο, είμαι τελευταία δύο λεπτά και εγώ. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σασόρη, τον συνάδελφο, καταρχάς πώς θα στο θέμα των περαιτέρω περικοπών στο επικουρικό ταμείο πρώτον και δεύτερον ε, όταν έχουμε να καταβάλουμε δύο ε, διαφορετικά ποσά ως εισφορά δική μας το παράρτημα επαριθμών τρία φορά, μόνο τους Ιταλούς και Γάλλους σε ένα βαθμό και τους ε, Λουξεμβουριούς συναδέλφους αλλά δεν εμφανίζονται και βλέπουμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε δύο ομάδες ποσών που καταβάλλονται επειδή κάποιες εθνικότητες βουλευτών θα είχαν ε, χαμηλότερη σύνταξη από κάποιες άλλες. Και βλέπουμε ότι οι Γάλλοι και οι Ιταλοί έχουν ένα σύστημα που τους επιτρέπει να συμπληρώσουν και μάλιστα πάνε πολύ περί, σε επίπεδο πολύ ψηλότερο από αυτό των εθνικών αντίστοιχων συντάξεων. Αυτό είναι ένα θέμα που δεν αφορά μόνο την επικουρική βέβαια σύνταξη, αλλά στην επικουρική 1500 ευρώ το χρόνο, το μήνα πληρώνει το κοινοβούλιο και τι έχουν και σε εθνικό επίπεδο δικαίωμα στη σύνταξη οι βουλευτές. Δηλαδή χρηματοδοτούνται δύο και τρεις φορές στις τάξεις αυτές. Ερωτώ λοιπόν. Έχετε κάποιο σχέδιο που μπορείτε να μας ανακοινώσετε. Έχουμε να κάνουμε πολλαπλά στεξιωτικά συστήματα και τελικά πάντα την πατάει ο Ευρωπαίος φορολογούμενος. Έχετε το λόγο. Και ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Για την κυρία Γιάλα πρώτα. Το Helpdesk. Ήταν μια επιθυμία της Επιτροπής σας για την ε, οργάνωση ενός τέτοιου helpdesk. Ε, αλλά πρέπει να σας πω ότι έχουμε διάφορα κέντρα που επεξεργάζονται το ίδιο θέμα της απαλλαγής. Έχουμε τη γραμματεία της Επιτροπής, έχουμε την επιστημονική υπηρεσία, ε, τους συνεργάτες. Δεν θέλουμε να θεσπίσουμε ένα επιπλέον ε, όργανο. Προσπαθούμε να συντονίσουμε μέσα από ένα helpdesk το οποίο είναι εγκατεστημένο στο Policy Department και έτσι συντονίσει τη δουλειά των διαφόρων φορέων και υπηρεσιών και ταυτόχρονα συνδυάζει όλη αυτή την πραγματογνωμοσύνη για να την προσφέρει μετά στους ενδιαφερόμενους. Επίσης, ρωτήσατε τι συνέχεια δίνει το Προεδρείο. Βεβαίως ε, ενημερώνεται για κάθε απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού το Προεδρείο, όπως άλλωστε και κάθε απόφαση οργάνων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο είναι σε τελική ανάλυση όργανο πολιτικό. Εγκρίνει και σε όρους πολιτικούς οποιαδήποτε τέτοια απόφαση. Άλλωστε και ο Αντιπρόεδρος κ. Σασόλεο νομίζω παρουσίασε πολύ εύγλωτα την κατάσταση και ότι μπορεί να προκύψουν διαφορετικές θέσεις ε, και αποφάσεις σε σχέση παραδείγματι με την καταποκοπή αποζημίωση ε, και εν τέλει με τις πλειοψηφίες του και τις μειοψηφίες του βεβαίως λαμβάνει τις αποφάσεις το Προεδρείο. για τους διαπιστευμένους βοηθούς. Έχει ενημερώθει το Προεδρείο ότι μέρος της ευθύνης, μεγάλο μέρος της ευθύνης το έχουν τα, ε, οι πολιτικές ομάδες και οι ίδιοι βουλευτές για στο να συμπληρωθεί η δεκαετία, ιδίως όταν λείπει ε, μικρό χρονικό διάστημα για να καλυφθεί η δεκαετία. Αλλά βεβαίως μπορεί και το Κοινοβούλιο να συμβάλλει εφόσον μπορεί ε, να αποφασιστεί ότι είναι απαραίτητη μια ad hoc διαδικασία και εφόσον βεβαίως είναι και η οι ε, ίδιοι ενδιαφερόμενοι, διατεθειμένοι να παραμείνουν μέχρι να συμπληρωθεί δεκαετία και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Κοινοβούλιο. Είχαμε ιδιαίτερα με την αλλαγή του συστήματος του 2009 πρόβλημα σε σχέση με τις συμβάσεις και κυρίως γιατί δεν είχαμε στη θέση μας όλα τα έγγραφα. Και αυτό έπαιξε το ρόλο του σε μια έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, ε, που έλεγξε το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού της ΠΕΡΣ γιατί δεν είχαμε τα στοιχεία για τη συμβάση της μας και τελικά το αποδείξαμε ότι όλοι αυτοί ήταν, ε, είχαν συμβάσεις. Ε, εξοπλισμός γραφείων των βουλευτών έχει αποφασιστεί από το Προεδρείο πως με τη νέα θητεία στις Βρυξέλλες για κάθε βουλευτή θα προβλέπεται η δυνατότητα να έχει δικό του γραφείο συν δύο γραφεία για τους συνεργάτες του, είτε είναι αυτοί οι ασκούμενοι, είτε είναι διαπιστευμένοι βοηθοί, κάτι το οποίο χρειάζεται οπωσδήποτε. Ε, μπορέσαμε λοιπόν να προβλέψουμε, χάρη στην ολοκλήρωση του κτηρίου Μάρτεν, στο οποίο έχουν μεταφερθεί χίλιοι εργαζόμενοι, ε, αποδεσμεύθηκε χώρος γραφείων που μπορεί να καλυφθεί από τους βουλευτές. Στο Στρασβούργο είναι πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση γιατί δεν θέλουμε να αγοράσουμε επιπλέον κτίριο ούτε και να μισθώσουμε επιπλέον κτίριο στο Στρασβούργο. Έτσι λοιπόν εδώ ε, το πρόσθετο δυναμικό θα δημιουργηθεί κατά τα δύο τρίτα των όσων ε, θα επιθυμούσαμε και στο πλαίσιο βέβαια της γενικής διαχείρισης ε, θα μοιραζόμαστε περισσότερους χώρους με κάποιες μικροπροσαρμογές βεβαίως και ως προς, το, προς την έκταση γραφείων, προς την επιφάνεια γραφείων που αντιστοιχεί στην Επιτροπή και το Συμβούλιο. Πάντως, δεδομένων των συνθήκων, θεωρήσαμε ότι ήταν σκόπιμο κάθε βουλευτής να έχει στο Στρασβούργο το δικό του γραφείο και ένα επιπλέον για το προσωπικό του. Και για να προστατευθεί βέβαια το απόρριτο και ο ιδιωτικός βίος, κρίθηκε αυτό απαραίτητο. Αυτή είναι η προσπάθειά μας τώρα και για αυτόν τον λόγο κάνουμε αυτή την προσπάθεια, όπως είπα. Αυτό καθίσατε δυνατό χάρη στον περιορισμό και τη παρουσία τη δίκη του Κοινοβουλίου στα δύο τρίτα. Για τον ε, κύριο Αλή, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τη θετική σα ε, αξιολόγηση, τη συνολική αξιολόγηση. Για τον οίκο τη Ευρωπαϊκή Ιστορία. 150.000 είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουμε για τους επισκέπτες. Τα πρώτα, θετικά, τα πρώτα αποτέλεσματα είναι θετικά, αλλά έχετε και δίκιο ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα ακόμα για να ενισχύσουμε τις ομάδες των επισκεπτών. Θα πρέπει να έχουμε στενότερη συνεργασία με τη Νέα Βουλή, ε, βουλευτές και βεβαίως ε, βοηθή των βουλευτών να μην το λησμονούν ε, αυτό, γιατί είναι μια, μεγάλη, μια πολύ καλή δυνατότητα που προσφέρεται στις ομάδες των επισκεπτών και των βουλευτών. Άλλωστε και τα γραφεία των αντιπροσωπιών, πρεσβείες και τα λοιπά μπορούν να δίνουν ε, τη δυνατότητα αυτή, μπορούν να αποστέλλονται λοιπόν ε, ε, επισκέπτες εκεί και υπάρχει ήδη στρατηγικό σχεδιασμός, πιστεύω πάντως ότι μπορούμε να βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο. μονάδα συμμόρφωσης στην νομοθεσία Regulatory Compliance Unit. Να σας δω λίγο το υπόβαθρο. Μέχρι τώρα είχαμε συζητήσει περιπτώσεις, ε, επιμέρους ζητήματα, προβλήματα, αλλά και καταχρήσεις σε διάφορες μονάδες. Αυτό που συνέβαινε λοιπόν ήταν ότι μπορεί να εστιάζαμε σε μια συγκεκριμένη μονάδα για να είμαστε απολύτως βίαιοι ότι ε, εξασφαλιζόταν το απόρριτο, η εμπιστευτικότητα ε, για να μην ε, πληγεί άδικα είτε υπάλληλο είτε βουλευτής. Όλα αυτά λοιπόν τώρα τα διαχειρίζεται μία μονάδα χωριστή, η οποία θα έχει και τη σχετική τεχνογνωσία, εμπειρογνωμοσύνη για να τα διαχειρίζεται καλύτερα. Όλη αυτή η εμπειρία λοιπόν συλλέγεται, βελτιώνεται, ήδη έχουμε πολυθετικό αντίκτυπο καταγράψει και πιστεύω ότι είμαστε στο δρόμο για τον κύριο Γιάβορ που μίλησε για τη γενική αποζημίωση, κατά αποκοπήν αποζημίωση γενικών εξόδων. Τοποθετήθηκε ήδη ο αντιπρόεδρο κύριο Σασόλη. Έχει ολοκληρώσει εργασίες της ειδική ε, ομάδα. Ο πρόεδρος ε, Καγιάννη έκανε τη σχετική διαπίστωση πως ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Επιτροπής αυτής στο Προεδρείο, το ανακοίνωσε. Άλλοι αισθάνονται ίσως πιο ικανοποιημένοι, άλλοι λιγότερο. Εν πάση περιπτώσει όμως ε, και με βάση την δημο... τις αρχές δημοκρατίας η ψηφοφορία έβγαλε το αποτέλεσμα που έβγαλε και οπωσδήποτε οι εργασίες θα πρέπει να συνεχιστούν κάποια στιγμή. Για την ε, απόδοση μη δαπανηθέντων ποσών Έχετε τη γραπτή πληροφορία, πιστεύω, λάβει στις γραπτές μας απαντήσεις. Όπως και για τον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό. 600 είναι βουλευτέ που έχουν μέχρι στιγμή καταθέσει στοιχεία ενό τέτοιου λογαριασμού, έχουν δηλώσει ένα τέτοιο ε, χωριστό λογαριασμό και έχει ενημερωθεί το Προεδρείο. ασφάλεια και το τι κάνουμε στον τομέα αυτών. Εδώ λοιπόν καταρχάς ανέλαβα την πρωτοβουλία ε, να προσκαλέσω ειδικού σε θέματα εκλογικών αναμετρήσεων από τα κράτη-μέλη για μια ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Έτσι λοιπόν ε, συνήλθαν σε μια κοινή συνάντηση, αντάλλαξαν εμπειρίες, βέλτιστες πρακτικές για την κυβερνοασφάλεια, ιδιαίτερα κατά την ε, εκλογική αναμέτρηση, για την εκλογική αναμέτρηση δεν σα ε, ξαφνιάζει φαντάζομαι αν σας πω ότι η Εσθονία διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό γιατί έχει και τη μεγάλη εμπειρία αλλά και είχαμε και σημαντική παρουσία ε, τσέχων ε, εκπροσώπων. Ε, εν πάση περιπτώσει όμως όλοι και όλα τα κράτη έχουν ε, λάβει τη σχετική ενθάρρυνση, ακόμα και αν δεν έχουν ε, πολύ προηγμένη τεχνογνωσία, να βελτιώσουν τι επιδόσει του ω προ την ε, προστασία, την προστασία για τι εκλογικέ αναμετρήσει. Fake news έχουμε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράσεω τη συνεργασία, γιατί έχει αναπτύξει εκεί μια εξαιρετική ποιότητα μονάδα και έτσι έχουμε μια συνεργασία με πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου και υποστήριξη και οικονομική ε, παρακολουθούμε στενότερα τις εκλογές, σε συνεργασία κατά την περίοδο των εκλογών και με, άλλα, με τα άλλα θεσμικά όργανα. Ε, και πιστεύω ότι είναι καλό να ενισχυθεί αυτή η δουλειά της σχετικής μονάδας υπηρεσίας εξωτερικής δράσης για όλους, για το καλό όλων πρέπει να συνεχιστεί και να ενισχυθεί. Και το νομοθετικό ίχνος ή αποτύπωμα με τον κύριο Ντεγιόνκο, ο οποίο έχει ιδιαίτερα αγωνιστεί για το θέμα αυτό με την έκθεσή του. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να παρακολουθούμε ε, αυτό πάντα σε εκούσια βάση γιατί είναι υποχρεωτικό το αποτύπωμα να καταγράφεται αυτό. Ο πρώτος στόχος λοιπόν της εξασφάλισης μιας δυνατότητας για την ε, ε, καταγραφή του ίχνους, του αποτυπώματος, νομίζω έχει πραγματοποιηθεί. Από εκεί και πέρα πρέπει και ο ίδιος ο βουλευτής να το εισαγάγει στον ιστότοπό του. Έχει γίνει σχετική ενημέρωση πως υπάρχει ένα εργαλείο της Transparency International και μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Έχει γίνει μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων στο Προεδρείο που έχει εντατικά ασχοληθεί με το θέμα της διαφάνειας και θα επαναλάβει τη συζήτηση αυτή σε ειδική σύνοδο, με ειδικό θέμα στη μερίσια διάταξη στο μέλλον. Ο κύριο Δε ρώτησε επίσης ε, σχετικά με την ε, επικοινωνιακή πολιτική και αν αυτή απευθύνεται μόνο σε νέους ή αν έχει ευρύτερο φάσμα αποδεκτών. Η απάντηση είναι ότι και χάρη στον προπολογισμό έχουμε μπορέσει να υποστηρίξουμε πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν τη δουλειά των πολιτικών κομμάτων, καθώς με αυτά μπορούμε να εξασφαλίσουμε την, τον όρο του πλουραλισμού, όλο το πολιτικό φάσμα λοιπόν μέσω των, πολιτικών, των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων που έτσι έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν σε διαφορετικές και συγκεκριμένες ομάδες αποδεκτών από το ίδιο το Κοινοβούλιο τώρα. Έχουν αναλυφθεί ε, διάφορες πρωτοβουλίες, ε, επίσης ευρέως φάσματος. Ο πρόεδρος Ταγιάννη, παραδείγματι, έχει ξεκινήσει και δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα τις τελευταίες εβδομάδες για το τι κάνει η Ευρώπη για μένα ένα πρόγραμμα που παρουσιάζει τις ε, αναφορές 100.000 διαφορετικών θέσεων, μονάδων, υπηρεσιών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό επίπεδο. Τι έχει κάνει η Ευρώπη για μένα σε διάφορα ζητήματα, σε διάφορα θέματα πρακτικά, όχι μόνο στην νομοθεσία, αλλά παραδείγματι τι, έχουμε, τι έχει προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους διαβητικούς, ε, αν μπορέσει να ενημερωθεί ο πολίτης ότι βοηθείται ο διαφητικός από κονδύλου του Ευρωπαϊκού πολίτης, ε, Προϋπολογισμού ε, ή ότι οι ποδοσφαιρόφιλοι έχουν επωφεληθεί από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό ή οτιδήποτε άλλο, τότε θα διαπιστώσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βελτιώνει τη ζωή μου για τον σκύλο επί παραδείγματι, που είναι ο σημαντικότερος σύντροφος για πολλούς από τους πολίτες μας αν παραδείγματι ενημερωθεί ότι να έχει διευκολυνθεί η δυνατότητα του σκύλου να συνοδεύει τον κύριο του στα ταξίδια του, ή οι ζωοτροφέ για σκύλου κτλ. έχουν βελτιωθεί χάρη στην νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε αποκτά ιδιαίτερη, αναγνωρίζεται η ιδιαίτερη εχουν βελτιωθει χαρη στην νόμο τη. Όλα αυτά λοιπόν σε έναν ιστότοπο με 2.000 περίπου ε, αναφορέ που υπάρχουν ε, μέσα σε μία σελίδα μόνο, με μια απλή γλώσσα, κατανοητή γλώσσα και πιστεύω ότι είναι ένα καλό ε, εργαλείο επικοινωνίας και ενημέρωση του πολίτη. Από το Δεκέμβριο ανοίγουμε την ε, application, την εφαρμογή τόσο σε Android όσο και σε Apple ε, πολίτης, την εφαρμογή πολίτης, αλλά επίσης προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε και τη διασύνδεση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και των τοπικών και περιφερειακών αρχών Ήδη είναι εκατοντάδε χιλιάδε οι πολίτε οι οποίοι το έχουν πράξει αυτό. Περί του 5.000 έχουν ιδιαίτερη δραστηριότητα. Έχουμε μάλιστα προσφέρει μια σειρά από προγράμματα εκπαιδευτικά κτλ. Για να καλύψουμε αυτό το θέμα. Ο κύριος Δεγιόν ρωτάει ακόμα για τον ε, οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Είχαν ε, λείψει τρεις υπάλληλοι και επιβαρύνθηκαν υπερβολικά οι υπόλοιποι τρεις. Ε, ήρθαμε λοιπόν ε, οι υπόλοιποι είχαν υποστεί σημαντική επιβάρυνση για υπερβολικό φόρτο εργασία. Μιλήσαμε με την αντίστοιχη επιχείρηση που του προσλαμβάνει και λάβαμε διαβεβαίωση πω θα τηρηθούν οι αρχέ και οι κανόνε του βελγικού δικαίου. Ο κύριο Γκερμπράντι ρώτησε για το στεξιωτικό ταμείο. Σωστέ είναι οι πληροφορίε σα. Πρόκειται για ένα πλάσμα δικαίου που ακολουθεί το ε, λουξεμβουριανό δικαίωμα, το δίκαιο του Λουξεμβουρού, η υποχρέωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι υποχρεώσεις του απορρέων πρώτον από το καθεστώς των βουλευτών του 2009, όπου έχει αναφερθεί ρητά η υπαγωγή του στεξιωτικού δικαιώματο στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, αλλά και απορρέει ταυτόχρονα από μια απόφαση του Προεδρείου πάλι του 2009, της 18ης συγκεκριμένα Μαρτίου του 2009 και της 1ης Απριλίου του 2009 και το ξέρω γιατί ήταν η πρώτη συνεδρία στην οποία συμμετέσχον ως Γενικός Γραμματέας και είχα τη μεγάλη χαρά να βρω το θέμα αυτό μπροστά μου να με περιμένει. Εκεί λοιπόν αναγνωρίζεται ρητά η νομική βάση όπως άλλωστε έχει συστήσει και η νομική υπηρεσία η οποία ωστόσο είχε επισημάνει ότι δεν μπορούσε πλέον να ε, πραγματοποιηθεί αδίποτε τροποποίηση. Τροποποίησης έφερε το Προεδρείο, οι οποίες έχουν επιβεβαιωθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Άρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα ως να, να λάβει ακόμα, να λαμβάνει και στο μέλλον αποφάσεις προς τους όρους προσφοράς της υπηρεσίας. ζητήματα τίθενται ως προς τα κεκτημένα δικαιώματα, τα acquired rights όπως λέγονται, δηλαδή μέλη του Ταμείου του εξοδοτικού που δεν έχουν ακόμα ε, βγει στη σύνταξη, γιατί επί παραδείγματι αυξήθηκε το όριο εξοδότηση στα 63, όπως ρητά έχει ε, εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ήταν νόμιμη αυτή η αύξηση στα 63 χρόνια, αλλά τίθεται το ζήτημα εάν ήταν εάν ε, εάν ε, υπάρχει παρέμβαση του Προεδρείου ως προς το σημείο εκείνης αυτών των θεμελιωθέντων, των θεμελιωμένων δικαιωμάτων. Αυτά και για τις ερωτήσεις τώρα της Προέδρου της Επιτροπής που θα μου τις υπενθυμίσει. Ναι, ήταν για τους Ιταλούς και Γάλλους βουλευτής. Λοιπόν, αυτό είναι βαρύδι του παρελθόντος, όταν δεν υπήρχε Ευρωπαϊκή Σύνταξη. Δεν όριζε δηλαδή το ε, καταστατικό των βουλευτών ε, Ευρωπαϊκή Σύνταξη και άρα είχαν τη δυνατότητα, το δικαίωμα τουλάχιστον για μια σύνταξη οι ευρωβουλευτές. Αυτό αφορούσε τους Γάλλους και Ιταλούς ευρωβουλευτές. Και εδώ υπάρχει μια συστηματική... Να, και τους Λουξεμβούργιους. Ε, άρα εδώ έπρεπε να γίνει η επιλογή και συστηματικά επιλεγόταν ε, το Σταξιδοτικό Ταμείο με επικουρική Ωστόσο, η υποχρέωση υπάρχει για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την έχει διαπιστώσει η νομική Υπηρεσία, πως απορρέει από το καταστατικό και την απόφαση του Προεδρείου του 2009, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να αλλάξουν οι όροι εκτέλεσης υποχρέωσης. Ο κύριος Σασόλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήδη απάντησε ο Γενικός Γραμματέας. Θέλω να πω ότι η άποψή μου είναι ότι οι κανόνες πρέπει πάντα να γίνονται σεβαστοί. Και ε, όσον αφορά το θέμα το συνταξιοδοτικό, εμείς δεν έχουμε διπλό ή τριπλό καθεστώς. Έχουμε ένα καθεστώς και έχουμε νομικές υποχρεώσεις που θα πρέπει να σεβαστούμε. Η έλλειψη σεβασμού αυτών των νομικών υποχρεώσεων θα οδηγούσε Βεβαίω σε προσφυγή στο δικαστήριο. Και αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε να συμβεί. Όσον αφορά την απόφαση της 4 η Νοεμβρίου του 1981 που αφορούσε την εξισορρόπηση των ευρωπαϊκών συνταξιών με εκείνους που δεν είχαν σύνταξη ήταν μια απόφαση που ακόμα αφορά 254 βουλευτές Ιταλός, 254 βουλευτές Γάλλους και τους Λουξεμβούργους που τότε ήταν σε αυτή την κατάσταση δεν είναι πλέον. Όσον αφορά την απόφαση για το συνταξιδοτικό ταμείο, όπως αναφέρθηκε, πρέπει να σεβαστούμε τους κανόνες και την απόφαση του Προεδρείου που ελήφθη το 2009, το 2024 θα πρέπει να συμμορφωθούμε στις υποχρεώσεις που αποφασίσαμε. Όχι εμείς, αυτούς πρέπει να σεβαστούμε την απόφαση του 2009, εκείνων που την πήραν. Μια παραβίαση αυτού θα οδηγούσε σε διαφορά και σε προσφυγή στο ΔΕΚ. Αυτό δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβεί. Είναι ένα και μοναδικό το συνταξιδοτικό καθεστώς αλλά υπάρχουν νομικές υποχρεώσεις που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να επιληθούν. Θα πρέπει να το σκεφτόμαστε εμείς κάθε φορά που λαμβάνουμε ε, αποφάσεις ότι αυτές έχουν συνέπειες και συνεπάγονται ευθύνε. Εν, εν τη αυτή περιπτώσει και βάρη τα οποία δύσκολα μπορούμε να αποφύγουμε. Λυπούμε διότι έφυγε ο συνάδελφος Γιάβορ. Ήθελα να του ζητήσω όσον αφορά την ερώτησή του, όσον αφορά τη μεταρρύθμιση των αποζημιώσεων, να πω ότι βρίσκομαι σε δύσκολη θέση να μιλώ με εκπροσώπους ομάδων στους οποίους εγώ έδωσα υποστήριξη, αλλά οι αντιπρόεδροι τους καταψήφισαν τελικά. Εγώ τους δικαιώσα και οι αντιπρόεδροι καταψήφισαν. Αυτή είναι μια πρόσκληση που απευθύνω σε όλους. Θα ήθελα να υπάρξει διάλογος μεταξύ αντιπροέδρων των πολιτικών ομάδων. Διαφορετικά, ίσως ε, οδηγηθούμε σε πολύ άσχημες έτσι καταστάσεις. Διότι στην Ολομέλεια η ομάδα ζήτησε πρωτοβουλίες και προφανώς οι αντιπροέδροι δεν επίστησαν ε, για αυτό το αίτημα που υπευλήθη. Δεν έχουμε από κατάσταση των ε, επιστροφή των ποσών. Δεν θα υπάρξει. Θα το συζητήσουμε στην επόμενη θητεία, αγαπητή κυρία Πρόεδρε, και πιθανότατα ελπίζω ότι οι διατάξεις που θα επανεξετάσουν τις υιοθετηθήσεις αποφάσεις με τις οποίες ήμουν αντίθετος θα επιτρέψουν να γίνει νέος υπολογισμός και αποκατάσταση αυτό, κάλυψη των δαπανών ε, κάτι που ζητήθηκε από το Κοινοβούλιο επανειλημμένα. Οι αντιπρόεδροι ψήφισαν διαφορετικά. Είναι όμορφη η δημοκρατία. Είναι όμορφη ακόμα και όταν χάνουμε για μια δίκαιη υπόθεση. Εδώ είναι πρόβλημα σοφιστίας. Να υπενθυμίσω ότι θα πρέπει να έχουν οι βουλευτές ε, μία επαφή και ένα διάλογο με τους αντιπροέδρους τους. Ευχαριστώ. Herr wünschen Κύριε Γκάλβιν, θέλετε να πάρετε ξανά το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα, για δύο θέματα μου επιτρέπετε. Θα ήθελα να συγχαρώ και να ε, ε, συμπληρώσω ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την ασφάλεια αλλά και για μια διαχείριση συνέχισης ε, συνέχεια των εργασιών στο Κοινοβούλιο για την ε, λειτουργία διαχείρισης κρίσεων και τις εξελίξεις και το σχεδιασμό για να μην υπάρχει διακοπή στη λειτουργία του Κοινοβουλίου, αλλά μια συνέχεια και μια συνάφεια στις διάφορες υπηρεσίες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, όσο προς την ασφάλεια. Και ένα δεύτερο σχόλιο θα ήθελα να συμφωνήσω απολύτως με την ερώτηση που έγινε για την κυβερνοασφάλεια και ο εσωτερικός έλεγχος θεωρεί ότι είναι από τους μεγαλύτερους κινδύνους που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και ο σχεδιασμός μας και ο προγραμματισμός μας ο ίδιος είναι να έχουμε πάντα παρουσία ε, στον έλεγχο και στην παρακολούθηση και τον εσωτερικό έλεγχο για τα όσα γίνονται για την Ιντερνετική ασφάλεια. Και τώρα ολοκληρώνουμε μια προκαταρκτική έρευνα που γίνεται. Πραγματικά οι δομές έχουν δημιουργηθεί ε, με τον επικεφαλής επόπτη της, των υπηρεσιών ασφαλείας και τις αντίστοιχε υπηρεσίες. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω, είναι πάρα πολύ σημαντική στη προτεραιότητα και σοβαρότατος κίνδυνος. Ο ένα Κίνδυνο που απειλεί το θεσμικό όργανο αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ε, Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ελπίζω οι διερμηνεί να μα δώσουν μερικά λεπτά ακόμα η συγκήτρια για να κλείσει. Α, με εκπλήσει που μου δίνετε το λόγο. Ε, ήταν καλή συζήτηση. Ε, είχα κι εγώ άλλες ερωτήσεις που δεν μπορούσα, μπόρεσα να κάνω. Ε, γιατί όταν απαντάτε τόσες πολλές ερωτήσεις με τόσο καλό τρόπο, τις 161, μία πάνω μία κάτω, δεν χάλεσε ο κόσμος. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, ήταν πολύ καλή η συνομιλία και νομίζω ότι θα πρέπει να παραμείνουμε σε επαφή. Αυτό ήταν το σύνθημα. Περιμένουμε ε, ε, μια προθεσμία για να δώσουμε τις ερωτήσεις μας. Ο κύριος Αλαφράκ έχει ζητήσει το λόγο, αλλά δεν τον είχα στον κατάλογο. Ε, πολύ σύντομα. Ναι, καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε χρόνο, απλώ θέλω να πω ότι έχουν γίνει μεγάλες πρόοδοι ε, στον τομέα της ασφαλείας και σε άλλες συζητήσει με το Γενικό Γραμματέα. Εθύμησα ότι ε, εγώ και άλλα δύο μέλη του Κοινοβουλίου πήραμε επιστολές βόμβες στο γραφείο μας. Ευτυχώς αυτό δεν επαναλήφθη μετά από τα μέτρα ασφαλείας. Για το Συνταξιδιωτικό ταμείο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα τελευταία ψηφίσματα ε, της έκθεσης Ρούμπικ και της απαλλαγής για τους Ιταλούς και τους ε, ε Γάλλους συναδέλφους ε, πρόκειται για 10,5 εκατομμύρια ετησίως. Και κάτι άλλο, κυρία Πρόεδρε, σημαντικό που σας ενδιαφέρει, που θα τα αφήσουμε για άλλη ευκαιρία για να μην ε, παρατείνουμε τη σημερινή συνεδρίαση. Πώς βλέπει ο Γενικός Γραμματέας και οι αντιπρόεδροι το θέμα των διορισμών. Όταν διορίστηκε ο Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχαμε μια απόφαση ε, που αφορά ε, τους διορισμούς των υψηλόβαθμων υπαλλήλων όλων των θεσμικών οργάνων. Αλλά αυτή είναι άλλη συζήτηση, κυρία Πρόεδρε. Ξέρω ότι μας ενδιαφέρει πολύ στην Επιτροπή μας και θα έχουμε σίγουρα την ευκαιρία να το δούμε σε μεγαλύτερο βάθος και λαμβάνοντας υπόψη πάντα την ε, προθυμία και τη διαθεσιμότητα του Γενικού Γραμματέα και των Αντιπρόεδρων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την κατανόηση ότι δεν μπορούμε τώρα πια να το συζητήσουμε αυτό. Πόσο μάλλον που στο Κοινοβούλιο ε, ε, η θέση του Γενικού Γραμματέα προκυρήστε. Το πρόβλημα νομίζω είναι στους Γενικούς Διευθυντές. <laughs> Θέλετε τώρα κύριε Γενικέ να αποπειραθείτε, να απαντήσετε. Γιατί ε, εδώ είμαστε το μαύρο πρόβατο, υπήν. Για το θέμα των διορισμών αυτό τον καιρό εκπονούμε κανόνες για να αναθεωρήσουμε τους παλιούς που ανάγονται το 2000 είναι περίπου 20 ε, ετών, 18 ετών. Ήταν ο προ, προκάτοχός μου. Ο πρόεδρος Σταγιάννη θέλει οι κανόνες αυτοί να ε, να προσαρμοστούν και με βάση την σημερινή διαδικασία. Δηλαδή προτείναμε από κοινού ε, να προτείνονται στο Προεδρείο περισσότεροι του ενός υποψηφί και ή δυνατόν πάντα να έχουμε εκπροσώπους άνδρες ή γυναίκες του υποεκπροσωπούμενου στην εκάστοτε περίπτωση. Και σε ερωτήσεις που είχαμε εδώ, ε, είχαμε συζητήσει σε προηγούμενες συζητήσεις ε, εκπροσώπους ε, θέματα της ακουρασόπησης γυναικών σε επίπεδο διευθυντών, γενικών διευθυντών. Τώρα έχουμε φτάσει στους τμήματάρχες. Όταν ήρθαν ήταν 23% οι γυναίκες τμήματάρχες και τώρα έχουν φτάσει περίπου στο 40%. Και ποια διαδικασία υλοποιούμε. Κάθε Γενικό Διευθυντή οφείλει να καταθέσει τρει προτάσει και στι τρει αυτέ προτάσει θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία γυναίκα. Και αν δεν υπάρχει τουλάχιστον μία γυναίκα, τότε επιφυλάσσομαι να ανοίξω το διαγωνισμό προς τα έξω για να έχουμε μια καλύτερη εκπροσώπηση. Άρα υπάρχει πάντα η δυνατότητα να διορίζονται γυναίκες που βεβαίως έχουν τα απαραίτητα προσόντα και έχουμε κάνει προόδους. Για τις διευθύντριες επίσης έχουμε κάνει πρόοδο στις γενικές διευθύντριες υπάρχει οπισθοδρόμηση μάλλον. Αυτή η αλλαγή ε, λοιπόν των κανόνων που ε, πρότεινε ο πρόεδρος έγινε δεκτή από το Προεδρείο, δηλαδή κάθε φορά ε, να έχουμε περισσότερες της μίας προτάσεις και υποψηφίους, όπως γίνεται με τους μηματάρχες και οι δυνατόν να έχουμε και τα δύο φύλλα. Αυτό είναι πολύ σημαντική πρόοδος, πιστεύω. Και ελπίζω και πριν τις εκλογές αυτό να επισημοποιηθεί και να ληφθεί και τυπικά η απόφαση στο Προεδρείο. Οπότε και εμείς ε, δείχνουμε επικοδομητική στάση στη συζήτηση αυτή και την ε, ε, Ασθενιζόμαστε και εμείς. Τελειώσαμε. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε όλοι και σας κύριε Γκάλβιν και σας κύριε Σασόρη και σας κύριε Γενικέ. Λέξη συνεδρίαση συνεχίζουμε αύριο σε 9 η ώρα το πρωί. Ευχαριστώ.